που υπάρχουν. Από τη μία έχουμε, παραδείγματο χάρη, την παγκοσμιοποίηση, έχουμε την ε, κακή αντιμετώπιση από τα μέσα ενημέρωσης ε, που οδηγεί σε κάποια δυσφορία. Η κρίση ή οι κρίσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι μεταξύ άλλων και η δημοκρατική νομιμοποίηση και η θεσμική κρίση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο πολίτης χάνει τις εξουσίες του. Επίσης βλέπουμε ότι θεσμοί που δεν είναι αιρετοί ή που δεν έχουν την πλειοψηφία παίρνουν μεγαλύτερη δύναμη και εξουσίες για να λαμβάνουν ε, κατεπίγουσες αποφάσεις ή για να ίσως θεσμοθετήσουν στο μέλλον και τις νέες αρχές. Ποιε είναι τώρα οι συνέπειες κατανομής που μπορεί να έχουν οι αποφάσει αυτών των μη ερετών φορέων για τους περισσότερους ανθρώπους. Το λιγότερο είναι ότι βλέπουμε πολιτικοποίηση πολύπλοκου ζητήματος, ε, όπως αυτό της χάραξης πολιτικής, και όλο και περισσότερες αμφισβητήσεις. Η καθιερωμένη προσέγγιση, μία από αυτές, σε ό,τι αφορά πάντα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, περιλαμβάνει την έννοια της ολοκλήρωσης μέσω διαβούλευσης. Αυτό σημαίνει ότι η λήψη αποφάσεων στο πολυεπίπεδο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δομικά, διαρθρωτικά πρέπει, θα έπρεπε να συνδέεται με τις απόψεις των πολιτών, τις εμπειρίες, τα βιώματά τους, και επίσης να περνάει από την πληροφόρηση, από την επικοινωνία και μέσω των ΜΜΕ. Άρα ε, ο σχηματισμός πολιτικής ε, γνώμης και της κοινή γνώμης σχετίζεται και με τη θεσμική λήψη αποφάσεων. In the EU, Τώρα, ολοκλήρωση μέσω δημοκρατικής διαβούλευσης. Αυτό το θέμα το έχουν ε, μελετήσει πολλοί ερευνητικοί όμιλοι, πολλές ερευνητικές ομάδες, και άλλοι φορείς, ιδίω στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου το ΡΕΚΟΝ, πώς θα αποκαταστήσουμε δημοκρατία στην Ευρώπη 2007-2011. με βάση ένα ιστοτό από το Όσλο και 20 εταίρους πέρυσι. Είχα το προνόμιο, όπως και ο Κρίστιαν Γιώργης, που είναι εδώ σήμερα, να μετα να συμμετάσχουμε σε, αυτή, σε αυτό το εγχείρημα. Θα μπορούσα λοιπόν τώρα να σας ε, πω το εξής. Η ολοκλήρωση μέσω της διαβούλευσης είναι όλο και ε, πιο επίκαιρη, ιδίως ε, τώρα, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη, τώρα που είμαστε σε περίοδο κρίσης. Και αυτό το αξίωμα θα σας το τεκμηριώσω αναφέροντας κάποιες παθογένειες του δημοκρατικού συστήματος σε συγκεκριμένα βήματα. Το πρώτο βήμα, σε ό,τι αφορά ε, την αποδυνάμωση των πολιτών, ε, την απώλεια της εξουσίας του πολίτη, σε ό,τι αφορά τη δυτή του ταυτότητα, ιδιότητα, ρόλο. Δηλαδή, ότι ο πολίτης αφενός είναι επίκοος ενός κράτους, μιας κρατικής εθνικής κοινωνίας, με κοινωνικο, οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα, από την άλλη πλευρά όμως είναι και πολίτης της Ένωσης ψηφίζει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που όμως περιθωριοποιείται όλο και περισσότερο παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Αποδυναμώνεται, είναι λιγότερο ορατό στη δημόσια σφαίρα για την πράσπιση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος ή ειδικότερα του συμφέροντος των πλέον ευάλωτων παραδείγματο χάρη, φορολογούμενοι, εν γέννη, μεσοαστική τάξη και ειδικότερα άνεργοι. Δυστυχώς βέβαια. Ποιες είναι οι διαβουλευτικές μέθοδοι για την ενίσχυση της συμμετοχής και της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι υπόσχονται σε σχέση ακριβώς με αυτή την κατάσταση της αποδυνάμωσης ε, των πολιτών ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά είναι εργαλεία για τη διόρθωση ορισμένων από, αυτό, από αυτές τις αδυναμίες και ανεπάρκειες και ιδίως αυτές που σχετίζονται με τις ασημέτριες ε, της ενημέρωσης και πληροφόρησης, την έλλειψη επικοινωνίας. Οι συνάδελφοι, όπως ο Νίμαν, έχουν συνεργαστεί στο αυτό το ρέκον και έκαναν ε, κάποιες δηλώσεις. Παραδείγματο χάρη ότι θα πρέπει η στρέβλωση να διορθωθεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες για πράγματα που τα αγνοούν. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρευλώσεις και οι οποίες τρευλώσεις είναι παράγωγο της χειραγώγησης των προτιμήσεων με την χρησιμοποίηση πολιτικών στρατηγικών όπως είναι η συμβολική πολιτική ή προϊόντα παράγωγα ε, γενικώ διεφθαρμένων πολιτικών σφαιρών. Πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτές τις παθογένειες Έχουμε μια εργαλειοθήκη η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, ιδίω στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την αποτυχία των ε, δημοψηφισμάτων της Γαλλίας και της Ολλανδίας ε, για τη σταγματική συνθήκη. Υπήρξαν ε, αρκετοί πειραματισμοί, παραδείγματο χάρη τα deliberative polls, δηλαδή ε, το, Euro, το ευρωβαρόμετρο και άλλες δημοσκοπήσεις, ξέρουμε ότι παρακολουθούν, αλλά δεν δίνουν στους πολίτες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για αυτούς αν θέλουν να λαμβάνουν ε, ε, στάσεις και τοποθετήσεις με τα λόγου γνώσεως. Και δεύτερον, κάποιες, κάποια συνέδρια συνένεσης των πολιτών Η αλληλεπιδράση των πολιτών δεν είναι βέβαια το αντικείμενο αυτής της ε, ακρόασης, αλλά και η απαραίτητη πληροφόρηση θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να φτάσουν σε συνένεση παρά τις διαφορετικές προτιμήσεις, απόψεις και συμφέροντά τους. Και τρίτον, η διαλογική εκπροσώπηση Έτσι μπορούν να προβάλλονται ανταγωνιστικές, διαφορετικές εμπειρίες, απόψεις, να αντιπαραβάλλονται μεταξύ τους και έτσι δημιουργείται μια καθολική δειγματοληψία που περιλαμβάνει τις απόψεις, τις διάφορες απόψεις της δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση όπου Υπάρχουν κανόνες, προϋποθέσεις που ε, μπορεί κανείς να τι αποκαλέσει δίκες. Ανάμεσα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, στο πλαίσιο τη συνθήκη τη Λισαβόνα, υπάρχει χώρο για την πρακτική εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της συνέλευσης, convention, για την μεταρρύθμιση της συνθήκης αντί της διακυβερνητικής συνέλευσης ως αναλλακτική λύση. Και εδώ δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη συνέλευση που έχει συγκροτηθεί μετά το Λάκεν 2002-2003 ε, υπό τον Ζεσκάρντε Όχι. Υπήρξαν πολλά κενά τα οποία αντιμετωπίστηκαν ε, μετά και την αποτυχία αυτής της συνέλευσης διότι οι πολίτες ερωτήθησαν ε, εκ των υστέρων. Ε, βρέθηκαν πρωτοτελεσμένου. Είχε ήδη εκπονηθεί το σχέδιο συνταγματική συνδίκης και την είχαν υπογράψει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Γιατί δεν επιτράπει στους πολίτες να εκπροσωπηθούν δίκαια και ακόμη και λιγότερο μορφωμένη. Υπάρχει ένα βιβλίο του Νίλ Κλίξτιν για το Euroclass. Convention or two conventions, they offered ample opportunities και γίνεται λόγο για αυτέ τι δύο συνελεύσει που τελικά πρόσφεραν ε, στις ελίτ και σε ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται και να δουλεύουν εδώ στι Βρυξέλλες ή τέλο πάντων ε, στο κοινοτικό πλαίσιο. Δόθηκε δυνατότητα λοιπόν σε αυτούς να επηρεάσουν, αλλά δεν ακούστηκε η άποψη του απλού κόσμου που αυτός πλήττεται και περισσότερο ή αφορά, αφοράται περισσότερο από τις αποφάσεις. Τώρα έρχομαι στο κοινοτικο πλαισιο δοθηκε δυνατοτητα λοιπον σε αυτου να επηρεασουν αλλα δεν ακουστηκε η αποψη του απλου κοσμου που αυτο πληττεται και περισσοτερο η αφορα αφοραται περισσοτερο απο τις αποφασεις τωρα ερχομαι στο αλλο θεμα τους ε, μη αιρετούς φορείς τα μη εκλεγμένα όργανα και κυρίως μου για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε όμως και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μη πλειοψηφική λοιπόν φορείς, μη ερετή. Είναι απαραίτητη, θα ήθελα να πω. Αυτά τα όργανα είναι απαραίτητα, γιατί μπορούν να διαφυλάξουν το κοινό συμφέρον από εκλεγμένες πλειοψηφίε που όμως μπορεί να επηρεάζονται από συγκεκριμένα συμφέροντα και περιορισμούς. What does deliberative, what... Οι διαβουλευτικές μέθοδοι τι προσφέρουν Και γιατί βλέπουμε με καχυποψία αυτούς τους οφορείς αυτά τα όργανα, διότι περιορίζουν την εθνική κυριαρχία. Που φαίνεται να είναι η φόρμουλα της ευρωπαϊκής επιτυχίας, τουλάχιστον για δύο αιώνες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από το 1951 και μετά η δημοκρατική αυτονομία και η εθνική κυριαρχία δεν όμως απαιτούν ακριβώς το να μην μπαίνουν στο πρώτο πλάνο αυτοί οι μη αυτά τα μη εκλεγμένα όργανα σε σχέση με ε, το, τους εθνικούς ερετούς άρχοντες. Εδώ πιστεύω ότι η δημοκρατική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει να συμφιλειωθεί η ένταση μεταξύ αφενός ε, του input legitimacy και αφετέρου του output legitimacy, δηλαδή νομιμοποίησης ε, εισφοράς, ε, συνεισφοράς και νομιμοποίησης αποτελέσματος. The concept I want to propose... Η Πρόεδρος, με συγχωρείτε, ήδη έχετε μιλήσει 15 λεπτά. Βέβαια, επειδή είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, ε, θα σας αφήσω να, συμμετα... να συνεχίσετε. accountable sovereignty. Ε, Η λεγόμενη υπεύθυνη ε, κυριαρχία ή υπόλογη κυριαρχία φαίνεται να είναι μια αντίφαση ουσιαστικά, αλλά περιλαμβάνει ε, α, αυτόνομους ανεξάρτητους φορείς που όμως πρέπει να είναι υπόλογοι. Πρέπει δηλαδή να λογοδοτούν για τη συλλογιστική που διέπει τι αποφάσεις που λαμβάνουν. Παραδείγματο χάρη, ο Μάριο Ντράγκη που είπε ότι θα πάει στην Bundestag. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα είδος ε, υπόλογης ε, κυριαρχίας ε, που μπορεί να συμβαίνει στα κρατημέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή της αρεσιμότητας ε, των όρων που επιβάλλονται στις χώρες τις μνημονιακές ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμών Σταθερότητας. Επίσης, ένα που πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατική αυτονομία, ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζοντας την κρίση με τον τρόπο που το κάνουμε. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η έννοια της ε, εθνικής κυριαρχίας και να συμπεριλάβει και την έννοια της λογοδοσίας, της ευθύνης, κάτι το οποίο απαιτεί διαβουλευτικές δημόσιες διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι και κλεισμένων των θυρών, ανοιχτά, δημόσια. Έχω και ένα τρίτο σημείο που αφορά τη διανομή, αν θέλετε, ε, την ε, κατανομή των αντιπαραθέσεων ε, που έχουν, στην περίπτωση της κρίσης παραδείγματος χάρη, έχουμε έντονα διανεμητικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, ούτε μπορεί να γίνει υπερεθνικό κοινωνικό κράτος, αλλά παρόλα αυτά λαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες θα αλλάξουν την διανεμητική ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών τάξεων, ομάδων, στρωμάτων των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Είναι να χρησιμοποιήσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση μέσω του άρθρου 9 της Συνδίκης Λισαβόνας, της Συνδίκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριζόντια κοινωνική ρήτρα. Το άρθρο 9 ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τον ορισμό και την υλοποίηση όλων των πολιτικών και των δράσεών τη, μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα έλεγα, τι απαιτήσει που σχετίζονται με την προώθηση υψηλού επίπεδου απασχόληση, εγγύηση τη επαρκού κοινωνική προστασία, καταπολέμηση, κατά του, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και υψηλά επίπεδα υγεία, εκπαίδευση και προστασία ανθρώπινη υγεία. Δείτε τη βάση αυτή της συνθήκης όταν θα πρέπει να έχετε υπόλογους την παραδείγματος το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. και τις διαπραγματεύσει που γίνονται με χώρες όπως η Ελλάδα κτλ. Αγαπητοί ευρωβουλευτές, η οριζόντια αυτή κοινωνική ρήτρα, αυτή η διάταξη, όπως και η συνέλευση, το convention που λέμε, περιμένουν προτού ε, έχουν αποτέλεσμα να υπάρξει η ανάλογη δράση, δηλαδή να υποβληθούν και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έχουμε νεοσυσταθέντα όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν νέε εξουσίες και σίγουρα η διαβουλευτική μέθοδος δεν θα μεγαλώσει την απόσταση της Ένωσης από τον πολίτη, αλλά θα την σμικρύνει. Τρεις εκκλήσει έχω να υποβάλω. Πρέπει να καταπολεμηθούν οι δημοκρατικές παθογένειες και να διορθωθούν. Με την ανάπτυξη πρώτα απ' όλα μια μεθόδου εργασίας μέθοδο εργασία θα μπορούσε να είναι η διαβούλευση. Ιδίω εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το κατεξοχήν ε, αντιπροσωπευτικό των πολιτών σώμα, ενδυνάμωση των πολιτών. Δεύτερον, οικοδόμηση υποδομών, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα κυρίαρχα κράτη υπόλογα, αλλά το ίδιο και τους ανεξάρτητους μη ερετούς φορείς και όργανα. Και επίσης κάποια συνέδρια που θα πρέπει να γίνονται με τους εμπλεκομένους φορούς, φορείς, ε, όπως στις μνημονιακές χώρες για παράδειγμα. Θα μπορούσαν ίσως αυτά τα συνέδρια, αυτές οι συνεδριάσεις ε, να ε, συμφιλιώσουν κάποια μέτρα κοινωνικά με οικονομικά για παράδειγμα ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, τον δόκτωρα Ανδρέας Γκρός, μέλος του Ελβετικού Κοινοβουλίου και βέβαια είναι και πρόεδρος του Σοσιαδημοκρατικής Ομάδας, συνάδελφός μου, πρόεδρος της Δημοκρατικής Ομάδας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει σε 15 λεπτά να κάνω κάτι ε, σχεδόν αδύνατον γιατί έχω ακούσει πολλές παρεξηγήσεις ε, για το τι στη άμεση δημοκρατία. Ορίστε, ορίστε, εντάξει, καλώς. Θέλω να ξεκινήσω με τον... Ε, ξεπεράσουμε αυτή την κατάχρηση των όρων. Και είναι και ευκαιρία να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί καμιά φορά έχει κανείς την εντύπωση ότι ζει σε κάποια οργολιανή εποχή ότι όπου χρησιμοποιούν όλοι τις ίδιες λέξεις αλλά σημαίνουν άλλα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ακριβείς. Για μένα λοιπόν ο ορισμός, τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να μετράμε αν θέλετε είναι αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Αν τα κοιτάξουμε λοιπόν αυτά τα κριτήρια, βλέπουμε πως η δημοκρατία πρέπει να είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία επιλογή. Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να είναι ελεύθεροι. Αλλά, βεβαίω πρέπει να αντιληφθούμε και το τι εστί ελευθερία ελευθερία δεν είναι μόνο η επιλογή μεταξύ πέψη και coca Είναι η δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς μαζί με τους άλλους μια κοινή βάση για τη ζωή του. Η ζωή δεν πρέπει να είναι μοίρα προκαθορισμένη. Σκεφτείτε πως οι άνθρωποι σήμερα α, αντιλαμβάνονται την δημοκρατία, τις πολιτείες στις οποίες α, πολιτεύονται ως κάτι διαφορετικό από μια ημαρμένη. Νομίζω ελάχιστη. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι πως ε, η δημοκρατία περιορίζεται στο εθνικό κράτος παρά το ότι οι πραγματικές επιδράσεις στην καθημερινή ζωή σήμερα προέρχονται από υπερεθνικές δομές. Γιατί η δημοκρατία είναι και μια υπόσχεση για να υπάρχει μια υπόσχεση για ένα δίκαιο μοίρασμα των ευκαιριών, των δυνατοτήτων. Το εθνικό κράτος δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει περισσότερο. Γιατί το έθνος κράτος χάνει την αυτονομία, αλλά δεν υπάρχει ένα αντιστάθμισμα στο υπερεθνικό επίπεδο. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια ηγεμονία των οικονομικών δυνάμεων για να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των ε, διαφόρων ε, συμφερόντων και υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να πω πως υπάρχει μία έννοια η οποία είναι βεβαίως πολύ ευρύτερη από το ε, μονοπόλιο της νόμιμης βίας, γιατί βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης των ε, συγκρούσεων, γιατί το να μειώνουμε τις συγκρούσεις στην βία είναι λάθος. Οι συγκρούσεις είναι μέσω κοινωνικής διδαχής Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται διαδικασίες και κανόνες οι οποίοι δεν θα καταλήγουν στη βία αλλά στην κατανόηση. Και αυτή είναι νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση και γι' αυτό χρειάζεται η έννοια του πολίτη, σιτουαγέν στα γαλλικά και όχι μπουρουσουά μια διάκριση που δεν υπάρχει στα αγγλικά. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι να μπορούν να επηρεάσουν την ζωή τους. Και τώρα όταν μιλάμε για την άμεση δημοκρατία, ίσως μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα στην επόμενη διαφάνεια, η δημοκρατία δεν είναι κάτι, η άμεση δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο θα αντικαταστήσει την αντιπροσωπευτική. Είναι ένα επιπλέον εργαλείο αντιπροσώπευσης το οποίο ε, αφαιρεί το μονοπόλιο από την ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και η άμεση δημοκρατία αφορά ζητήματα και όχι πρόσωπα γιατί το, η λογική ενός συγκεκριμένου ζητήματος αμεσοδημοκρατικού είναι τελείως διαφορετική από το να εκλέξουμε ένα άτομο. Το να εκλέξουμε δηλαδή τον πρόεδρο της Κομισιόν δεν είναι άμεση δημοκρατία. Εντάξει, διευρύνεται η εκπροσώπηση οπωσδήποτε, αλλά δεν έχει σχέση με την άμεση δημοκρατία. Μπορώ να εμβαθύνω εάν θέλετε αναφέρομαι κύριο το δημοψήφισμα βεβαίως δεν είναι πάντα το ίδιο. Δεν είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι τελείως διαφορετικό τι εννοούμε από το εάν το προξενεί η κυβέρνηση ή ο λαός. Γιατί όταν το συζητάμε στην Ναπολεόντια παράδοση, κατά κανόνα χρησιμοποιείται και από δικτάτορες και δεν έχει ούτε μία σχέση μετά με τη δημοκρατία. Και το ε, βασικό σημείο θα έλεγα είναι πως η άμεση δημοκρατία είναι μια συνεισφορά στην δημοκρατία και βεβαίω είναι μια συνεχή διαδικασία. Ποτέ δεν θα φτάσουμε στην τέλεια δημοκρατία. Αλλά πάντα βεβαίω υπάρχει μια αφετηρία στη διαδικασία αυτή εκδημοκρατισμού. Και βεβαίω αυτό το οποίο είναι πιθανό το σημαντικότερο και το πιο πιστικό αλλά και δύσκολο μας δείχνει πως σήμερα έχουμε την εντύπωση πως ε, στην ε, πλευρά της πολιτείας έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο δεν ε, επιτρέπει στις κοινωνίες να εγκαταλειφθούν το δυναμικό το οποίο έχουν. Οι πολίτες θεωρούν ότι τους υποτιμούν οι πολιτικοί. Αν δείτε τα άτομα, αν δείτε το σύστημα, μπορούμε να πούμε πως ο σημερινός σχεδιασμός της πολιτικής αυτή η μείωση στο εθνικό κράτος, αυτή η μείωση στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία η ενδυνάμωση των μη ερετών ε, σωμάτων μας δείχνει την μη οργάνωση της κοινωνίας για να εκμεταλλευτεί πλήρως το δυναμικό της. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η απογοήτευση και τόσο κόσμος γυρνάει την πλάτη του στην πολιτική. Για να ξεκινήσουμε τώρα με το σχέδιο, αν θέλετε, ένα σχεδιασμό τη άμεση δημοκρατία. Το βασικό είναι λοιπόν πώ σχεδιάζουμε κάτι τέτοιο. Ήδη ο κύριο Σίλε και άλλοι σήμερα το πρωί είπαν πω ε, μια κακοσχεδιασμένη άμεση δημοκρατία είναι χειρότερη από το τίποτα. Γιατί? Γιατί έτσι χάνει και την αξιοπιστία η διαδικασία. Αν είναι τόσο άσχημα σχεδιασμένη. Αλλά όταν τη σχεδιάζουμε κατά τον τρόπο ώστε ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί, τότε έχουμε αυτό ακριβώς το οποίο λείπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω. Και απαρίθμησα κάποια στοιχεία. Βεβαίως η νομιμοποίηση είναι σαφής και θα έλεγα επίσης πως σε καιρό που υπάρχει, το, υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα με, την, με τα αποτελέσματα, θα θέλαμε ίσως λίγο περισσότερη διαδικασία και συνεισφορά. Οπότε, όταν προσκαλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν και αυτοί, αισθάνονται τμήμα μιας ευρύτερης διαδικασίας, υπάρχει και ταύτιση και βεβαίως και ενσωμάτωση. Ο καλύτερος τρόπος να τεθεί αυτό είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντίρενματ, ένας από τους μεγάλους Ελβετούς συγγραφείς. Είπε πως οι Ελβετοί, όπως είπε ο Γκέραρτ το πρωί, ήταν πολύ διαφορετικοί, δεν είχαν κοινή ιστορία, κοινή γλώσσα, κοινό πεπρωμένο, κοινή θρησκεία. Το μόνο το οποίο έχουμε κοινό, είχε πει ο Ντίρενματ, είναι λοιπόν πως οι Ελβετοί έχουν την ευκαιρία κάθε τέσσερις μήνες να συζητήσουν τις διαφορές τους και οι αποφάσεις λαμβάνονται σεβόμενοι αυτές τις διαφορές και με τη συμμετοχή των ανθρώπων. Γιατί βεβαίως γίνεται σεβαστή η διαφορετικότητα, πάντα έχει ο καθένας μία ενότητα βεβαίως, αλλά ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ε, δει αυτή την ενότητα σε ένα άλλο επίπεδο. Υπάρχει τεράστια συζήτηση, επικοινωνία, που η επικοινωνία είναι και αν θέλετε η πηγή της άμεσης δημοκρατίας και έτσι δημιουργεί κανείς δημόσιες σφαίρες. Όχι μόνο μία, αναρρύθμιτες, εκατοντάδες χιλιάδες, όπου ο κόσμος ε, συναντάται, συζητά, άλλοι ακούνε, γενικώ υπάρχει συμμετοχή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Διότι υπάρχουν διάλογοι ε, βάση του αντικειμένου όταν επιλέγονται κάποιοι οι οποίοι θα συζητήσουν. Το 19ο αιώνα είχαμε και ένα κίνημα που αγωνίστηκε για την άμεση δημοκρατία στην Ελβετία ε, σε μια εποχή που ούτε φωτογραφίες υπήρχαν. Φυσικά δεν μιλάω καν για τηλεόραση, κινηματογράφο ή επικοινωνιολόγους κτλ. Το πιο δύσκολο είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβει κάποιος γιατί μετά τις εκλογές ε, με τις εκλογές μάλλον, γιατί μετά τις εκλογές μπορείς να δεις αν αυτός ε, τηρεί αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Και φυσικά και η λογική βοηθάει στη συζήτηση και στην κατανόηση. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης συμβάλλει στην ε, διασαφήνιση των ενιών είναι το εξής. Όπως είπα αρχικά, ε, παίρνει αυτό που σου λέει περισσότερο. Δημιουργείς όμως και αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο. Κοινότητες, κοινωνίες, διότι δεν μπορεί κανείς ε, να αποκτήσει κοινωνίες και κοινότητες αν δεν ενεργοποιηθεί ο κόσμος. Η ταυτότητα είναι το αποτέλεσμα κοινή δράσης. Γιατί όταν κάποιος είναι παθητικός, χάνει την ταυτότητά του. Το ίδιο γίνεται και με τις κοινότητες. Αν υπάρχει αίσθηση του ανήκειν, ε, αν υπάρχει διασύνδεση, μπορεί κανείς να δράσει ο σύνολο και να βιώσει κάτι ο σύνολο. Και το δεύτερο φυσικά είναι η έννοια του χάμπερ μας. Αλλά για την υλοποίηση αυτής της ε, συμμετοχής δημιουργείται η προϋπόθεση της συμμετοχής. Ε, η διαδικασία δημιουργεί τη συνθήκη, δημιουργεί τη διαδικασία. Τους Δήμους που μας λείπουν μπορούμε να τους αποκτήσουμε μόνο να προσπαθήσουμε να τους φτιάξουμε. Αυτό θα πει η άμεση δημοκρατία και δεν μπορεί κανείς να την μάθει. Δεν μπορεί να μάθει κανείς να κολυμπάει στην ξηρά, πρέπει να μπει στο νερό. Έτσι πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αν κάποιος δεν έχει επαρκή γνώση, του ζητάς να συμμετάσχει και αποκτά τη γνώση που του λείπει, αποκτά και ενδιαφέρον. Αν τον αφήνεις απ' έξω όμως, γιατί να τον ενδιαφέρει τίποτα. Όταν δημιουργούμε λοιπόν θεσμούς όπου επιτρέπουμε σε μικρό αριθμό ανθρώπων να αποφασίζουν για τους υπόλοιπους, δημιουργούμε διαδικασίες, ε, κίνητρα. Τελικά όλοι έχουν ε, το κίνητρο να ε, συζητήσουν μόνο όταν συναποφασίζουν όλοι και όχι λίγοι. Αυτέ λοιπόν οι λεγόμενε agenda initiatives, αυτέ οι πρωτοβουλίε για τη δημιουργία τη μέτσια διάταξη, του θεματολογίου και γενικότερα οι πρωτοβουλίε των πολιτών μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβάλλουν και τη δεξαγωγή ενό διαλόγου στην κοινωνία που μπορεί κάποιοι στην κοινωνία να μην την θέλουν αυτή τη συζήτηση, αυτό το διάλογο. Ο διάλογο όμω σίγουρα είναι η προπόθεση, όχι όμω και η εγγύηση τη αλλαγή. Αλλά αν κάτι δεν μπορεί καν να συζητηθεί γιατί αποκλείονται κάποια θέματα, τότε ποτέ δεν μπορεί κανεί να ε, πετύχει κάτι. Δημόσιε σφαίρες, λοιπόν, λείπουν, αποκτώνται με τη συμμετοχή. Το είδαμε και κατά τον παρελθόν με τους Ιρλανδούς και τους Δανούς που αποφάσισαν. Γιατί άρχισαν όλοι να ασχολούνται μαζί τους για να βλέπουν πώς αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Και άρχισαν να αποφασίζουν και οι άλλοι. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι μπορεί κανείς έτσι να δημιουργήσει δημόσιες σφαίρες. Όχι ότι όλοι θα κοιτάνε την ίδια τηλεόραση και θα διαβάζουν την ίδια εφημερίδα, αλλά ότι σε όλες τις τηλεοράσεις και σε όλες τις εφημερίδες θα επανέρχονται στην μέση διάταξη πιο πολύ ευρωπαϊκά θέματα. Τώρα, αν δεν κάνει το σχεδιασμό, τι πρέπει να προσέξει. Ποια στοιχεία του σχεδιασμού του μοντέλου θα αποφασίσουν ποιες είναι οι ανάγκες και τι θα χρειαστεί, τι θα βοηθήσει. Θα πρέπει να βοηθήσουν να έχουμε υπόψη μας πέντε κεντρικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι η είσοδος, η πόρτα από την οποία πρέπει κανείς να περάσει για να κινητοποιήσει, για να ενεργοποιήσει, να δρομολογήσει αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να είναι το 3%. Στη Ζηρίχη, ε, στο καντόνι αυτό, ε, ήμουν πάρα πολύ δραστήριος, είχαμε λιγότερο το 1%. Εντάξει, ίσως να είναι λίγο υπερβολικό. Έτσι θα έλεγε ο κύριο Γκέσνερ. Στην Καλιφόρνια είναι 5% πύχη. Ε, κάπου ενδιάμεσα. Όχι πάνω από 5 όμω, σε καμία περίπτωση. Γιατί, και αυτό το είπε και ο κύριο Μπρόν πριν. Όταν έχεις ένα μέσο που μόνο οι ισχυροί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, χάνεται η ομορφιά αυτού του εργαλείου, αυτού του μέσου, το οποίο δημιουργήθηκε, χάρη, δημιουργήθηκε στην γαλλική και ε, επανάσταση και μεταλαμπατεύτηκε μετά σε κάποιες άλλες χώρες. Πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο που να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτοί που δεν έχουν πολύ εξουσία, αλλιώς δεν έχει νόημα. αυτοί που έχουν την εξουσία φυσικά και δεν θέλουν να, υπάρχει ένα αντίβαρο, αλλά δεν μπορεί να περιμένει κανείς να έρχονται όλα από τους ισχυρούς. Οι ισχυροί δεν πρέπει να νιώθουν ότι είναι ασφαλείς, πρέπει να νιώθουν ότι μπορεί να χάσουν αυτή την εξουσία. Με παθητική στάση δεν πετυχαίνει κανείς τίποτε. Το δεύτερο μπορεί να μας το διδάξουν οι Ιταλοί, όχι μόνο όμως. Η όλη ιστορία της Βαϊμάρης μας το διδάσκει. Αν υπάρχει συμμετοχή, αν υπάρχουν κάποιες απαιτήσει έγκρισης, αυτό είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να υπάρξει μη επικοινωνία και μη ε, αποδοχή. Αν δεν υπάρξει επικοινωνία, πώς θα υπάρξει ενημέρωση. Στο ποδόσφαιρο το γκολ μπαίνει από το φάουλ, όχι από την κόκκινη κάρτα. Το γκολ μπορείς να το βάλεις αν έχεις κερδίσει ένα φάουλ και αν έχεις αποβληθεί. Ακούσαμε για την Ιταλία, ακούσαμε ότι οι μισές αποφάσεις ε, ήταν άκυρες. Για τον Περλουσκόνη έλεγε μείνετε σπίτι για να μην υπάρχει συμμετοχή του 50%. Οπότε ήταν άσκοπα όλα αυτά τα δημοψηφίσματα. Επίσης μπορεί κανείς να συγκρίνει το ευρωπαϊκό με το αμερικανικό σύστημα. Η διαπαφή, η διασύνδεση μεταξύ της άμεσης και της έμεσης δημοκρατίας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Δεν πρέπει να υπάρχει αντίθεση η αντιπαράθεση. Χρειάζεται συνεργασία, δεν χρειάζεται ανταγωνισμός. Γι' αυτό στα ελβετικά καντόνια υπάρχει η καλύτερη δυνατή συμμετρία. Από την έννοια ότι όταν το κοινοβούλιο ε, νομοθετεί, οι πολίτε όχι μόνο καλούνται να πούνε ή όχι, αλλά ακόμη και να προτείνουν, να κάνουν μια αντιπρόταση. μέσω της δικής τους πρωτοβουλίας και έπειτα γιατί προτείνει κάτι σε σχέση με αυτήν την πρωτοβουλία το Κοινοβούλιο. Και έχουν τρεις επιλογές ε, μετά οι πολίτες ε, να επιλέξουμε μεταξύ του τίποτα, α ή β. Τέταρτο στοιχείο. Υποτιμάται και αυτό πολύ. Πρέπει να έχουμε μια άλλη έννοια του χρόνου. Όχι του οικονομικού χρόνου. Διότι όσο ταχύτερα πρέπει κάτι να γίνει, τόσο πιο αποκλειστικά ή ε, μάλλον εξαιρετικά θα γίνει, δηλαδή αφήνοντα εκτό πολλού. Εμείς όμως το αντίθετο θέλουμε, να είναι ω το δυνατόν περισσότεροι εντός και όχι εκτός. Άρα θέλουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουμε ε, ταχυφαγία και πρόχειρε γρήγορε λύσει στο πόδι. Γι' αυτό μιλάμε για τρία-τέσσερα χρόνια. Διαδικασίε τριετή, τετραετή. Πρέπει να αλλάξει η έννοια του χρόνου λοιπόν. Και πρέπει να δούμε ποια είναι η έκβαση αυτή της, αυτής της πρωτοβουλίας. Αν κάποιοι κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, ίσως αλλάξουν άποψη, ίσω μορφώσουν άποψη, ίσως δηλαδή η θέση ε, που θα, θα προκύψει θα είναι διαφορετική από αυτή που κανεί θα νόμιζε. Χρειάζεται δικαιοσύνη, χρειάζονται κανόνες ε, και ευκαιρίες. Παραδείγματο χάρη. Κάποια κουπόνια για ταξίδια, συνεδριάσεις, για μεταφράσεις. Μπορούν να δώσουν δυνατότητα και σε πιο φτωχέ, αν θέλετε, οργανώσει να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να μην δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα είναι προνόμιο των ισχυρών. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. 20 λεπτά χρειάστηκε για να σας πω πράγματα που συνήθως μου χρειάζεται μισός χρόνος για να τα εξηγήσω. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε μπορούμε να επεκταθούμε στη συζήτηση περισσότερο. Ο προ... Η πρόεδρος, ναι βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι βέβαιη ότι αποτελέσετε πηγή έμπνευση για όλους μας. Και είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις και σχόλια. Όχι μόνο από εμάς τους δύο, αλλά έχουν έρθει και άλλοι συνάδελφοι. Συνάδελφος Μπρόνς είναι εδώ. Ξέρετε ότι έφυγε μια αντιπροσωπεία τη Επιτροπή ΑΦΚΟ με τον Καζίνη, τον πρόεδρό μα, για το Παρίσι εξού και δεν είναι παρόντα πολλά από τα μέλη τη Επιτροπή μα. Σα ευχαριστώ λοιπόν γιατί μα δώσατε πολύ τροφή για σκέψη. Τώρα να παρουσιάσω με πολύ μεγάλη χαρά την επόμενη ομιλήτρια, την δόκτωρα Νάντια Μπράουν Μπίντερ από την Ακαδημία Διοικητικών Επιστημών από το Σπάιερ. Καλώς ορίσατε. Μπορείτε και εσείς να μιλήσετε για 20 λεπτά, θα έχετε ίδια μεταχείριση με τους υπολείπους και μετά θα έχουμε και εμείς δυνατότητα να συζητήσουμε. Επίσης έχουν έρθει και κάποιοι από τους πρωινούς ομιλητές για να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου να σας μιλάω σήμερα. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω κάποια λόγια για μένα. Είμαι Ελβετίδα υπήκος και εργάστηκα στην νομική υπηρεσία, ήμουν νομικός σύμβουλος της ε, Ελβετικής ε, Συνομοσπονδίας και είχα ασχοληθεί με τις ε, διοργανώσεις δημοψηφισμάτων και πρωτοβουλειών πολιτών και με αυτή την ιδιότητα ή την πρώην ιδιότητά μου σας μιλάω σήμερα εδώ και ένα χρόνο ε, είμαι στην Γερμανία στο Πανεπιστήμιο του Σπάιερ όπως ακούσαμε τα κλασικά μέσα της άμεσης δημοκρατίας ήδη αναφέρθηκαν έχουμε την ε, πρωτοβουλία των πολιτών τα προαιρετικά δημοψηφίσματα και βεβαίως τα ε, παραδοσιακά δημοψήφισματα. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται σε διάφορα κράτη και στην Ελβετία τώρα ανεξαρτήτως των διαφόρων κατηγοριών κρατών. Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται και συζητούνται και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αυτονόητο είναι και σημαντικό είναι να το πούμε αυτό πως δεν μπορούν αυτομάτως να μεταφερθούν αυτά τα μέσα στο υπερεθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά είμαι πεπισμένη πώς οι ε, εμπειρίες εδώ πέρα μπορούν να μας βοηθήσουν. Εμπειρίες από την πράξη. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ελβετική διαδικασία για να δώσω κάποια παραδείγματα το τι σημαίνει δηλαδή να ζει κανείς σε μια χώρα σε μια χώρα η οποία ασκεί την άμεση δημοκρατία. Θα αναφερθώ τώρα στην εμπειρία από την πλευρά της διοίκησης όσον αφορά την διαχείριση και τη διοργάνωση δημοψηφισμάτων. Το πρώτο παράδειγμα είναι τα λεγόμενα δημοψίσματα τα οποία προκαλεί ο πολίτης με τη συλλογή 50.000 υπογραφών, αυτά τα οποία ονομάζουμε προαιρετικά. Τι συμβαίνει τώρα με τις 50.000 αυτές υπογραφές. Η νομική υπηρεσία του κράτους, το νομικό συμβούλιο του κράτους, εξετάζει τις υπογραφές και βεβαίως εξετάζουμε δύο πτυχές, εξετάζουμε το εάν οι Δήμοι έχουν κάνει σωστά την δουλειά τους οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσει την κάθε υπογραφή, πως ε, αυτός ο οποίος υπογράφει είναι ο ίδιος και πως έχει δικαίωμα ψήφου και δεν, έχει, δεν το έχει στερηθεί και δεν έχει υπογράψει δύο φορές την ίδια πρωτοβουλία. Ο δεύτερος έλεγχος αφορά την δεύτερη διάσταση θα λέγαμε, εξετάζουμε δηλαδή το εάν ένα άτομο έχει εγγραφεί και υπογράψει σε δύο διαφορετικούς δήμους. Δηλαδή μπορεί κατά τη διάρκεια της ε, προθεσμίας να μετακομίσει κάποιος και να μην μπορεί να το παρακολουθήσει ο Δήμος αν έχει υπογράψει ήδη κάπου αλλού. Εκεί είναι λοιπόν ένας δεύτερος έλεγχος. Μετά από αυτόν τον έλεγχο ξαναμετράμε τις υπογραφές. Μπορεί κάποιες να μην θεωρούνται έγκυρες είναι απλά τα πράγματα, αλλά αν είναι μέχρι και 7 υπογραφές κάτω από τις 50.000 ε, ε, τότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα χρειάζεται άλλη μια ανεξάρτητη καταμέτρηση κάτι το οποίο ούτως ή άλλως όμως συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια ούτως ή άλλως ε, πρέπει να γίνουν αυτές τις χθες πάρα πολύ γρήγορα υπάρχει μεγάλη χρονική πίεση, οπότε υποβάλλεται η πρόταση για ε, ένα δημοψήφισμα και θα πρέπει όλη αυτή η έλεγχη να γίνει συνήθως εντό ενός Σαββατοκύριακου γιατί ε, μπορεί να οδηγηθούμε από το προαιρετικό αυτό δημοψήφισμα σε δημοψήφισμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε έναν νόμο, σε να καταληφθεί ένα νόμο. Και βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Το δεύτερο παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το πώς ξεκινάει μια πρωτοβουλία πολιτών. Σε μια πρωτοβουλία πολιτών μπορούμε να ζητήσουμε την συμπλήρωση είτε την αλλαγή του συντάγματος είτε μέσω της διαγραφής είτε μέσω μιας πρότασης συγκεκριμένης διατύπωσης. Βεβαίως πρέπει και πάλι να δώσουμε βάρος στη διοικητική πλευρά το κείμενο βεβαίως της πρωτοβουλίας το συντάσσουν οι ενδιαφερόμενοι, όχι οι αρχές. Το κείμενο πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει η υπηρεσία, η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας γιατί βεβαίως ε, μπορεί να οδηγήσει το κείμενο αυτό να γίνει κατά λέξη συνταγματικό κείμενο και αντιλαμβάνεστε πως όλες οι επίσημες γλώσσες έχουν την ίδια ισχύ. Οπότε πρέπει να μην υπάρχει καμία διαφορά και στην ερμηνεία μεταξύ της γαλλικής, της γερμανικής ή της ιταλικής γλώσσας και εκδοχής του κειμένου. Η διατύπωση του κειμένου της ε, πρωτοβουλίας, όπως είπαμε βεβαίω, ανήκει στους ενδιαφερόμενους και όχι στις αρχές. Στην πράξη όμως, οι ενδιαφερόμενοι έχουν μια καλή ιδέα για το τι θέλουν, αλλά ξαφνικά όταν πρόκειται να γράψουν ένα άρθρο του συντάγματος δεν είναι και τόσο σίγουροι για το τι μορφή θα πρέπει να έχει. Γι' αυτό προκύπτει το ότι ζητάνε την βοήθεια των αρχών, μήπως θα μπορούσαν οι αρχές να κάνουν μια σύσταση. Αυτό είναι κάτι το λεπτό και ευαίσθητο. Οι αρχές και είμαι επευσμένη γι' αυτό. Και έτσι είναι και ο κώδικας, δεν μπορούν να κάνουν καμία σύσταση ούτε και απολύτως ουδέτερη. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί ποτέ η εντύπωση πως οι δημόσιες αρχές ε, επηρεάζουν την διατύπωση του κειμένου μιας πρωτοβουλίας. Αυτό το οποίο βεβαίως μπορεί να κάνει η δημόσια αρχή είναι να δώσει κάποια τυπικά κάποιες τυπικές συμβουλές, αν θα είναι λατινικά ή αραβικά τα νούμερα, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Αλλά επί της ουσίας ε, και του περιεχομένου δεν επιτρέπεται να βοηθήσει η υπηρεσία μας. Και βεβαίως χρειάζεται και ένας τίτλος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακαθόδες ορισμένες φορές γιατί η ο τίτλος της πρωτοβουλίας βεβαίως είναι ο τίτλος και της, ε, του δημοψηφίσματος. Αυτολεξή. Οπότε και αυτό το κάνουν οι ενδιαφερόμενοι και όχι η αρχή. Η αρχή πρέπει απλά να ελέγξει πως δεν είναι παραπλανητικός ο τίτλος, ότι δεν είναι διαφημιστικός, ούτε καν έμεσα ε, διαφημιστικός και βεβαίως ελέγχει η αρχή μας ε, πως ε, ο τίτλος δεν πρέπει να συγχαίεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ήδη τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα κριτήρια που σας ε, ανέφερα αφορούν την πρωτοβουλία και αυτά ελέγχονται από την καγκελαρία η οποία ελέγχει όλα αυτά τα κριτήρια η Επιτροπή σε τελική ανάλυση ε, πρέπει να καταθέσει μια πρόταση και τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, δεν μπορούν να καταθέσουν εκ των υστέρων αλλαγές και η πρωτοβουλία Εφόσον είναι επιτυχής, ε, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα την πρωτοβουλία αυτή να την αποσύρει. Και ε, βεβαίως ε, πρέπει να είναι γνωστό ποιος μπορεί να αποσύρει αυτή την πρόταση και ποια ακριβώς θα είναι τελικά η ε, πλειοψηφία. Αυτά λοιπόν είναι τα βήματα τα οποία καλείται να ελέγξει η νομική υπηρεσία του κράτους. Όλα αυτά τα καθορίζει μέσα σε ένα βούλευμα και αν αυτό το ε, βούλευμα δημοσιευτεί στις επίσημες γλώσσες, αυτομάτως αυτό ε, αποτελεί και το εναρκτήριο λάκτισμα για την συλλογή υπογραφών. Έρχομαι τώρα στο τρίτο παράδειγμα, το οποίο θέλω να σας παρουσιάσω. Πρόκειται για την ε, προετοιμασία της, ε, του δημοψηφίσματος. Και εδώ λοιπόν η υπηρεσία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, κυρίως ε, όταν πρόκειται να ενημερωθούν οι ψηφοφόροι. Έχουμε ακούσει λοιπόν επανειλημμένα σήμερα ότι η ενημέρωση είναι ένα σημαντικό στοιχείο, πρέπει να είναι ισορροπημένη, να είναι ουσιαστική και πρέπει να επιτρέπει στους ε, ψηφοφόρους να σχηματίσουν άποψη και να λάβουν απόφαση. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι πρέπει να πρόκειται για ε, αντικειμενικές ε, πληροφορίες και όχι για προπαγάνδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στην Ελβετία ε, πριν από ε, τις ε, πληροφορίες που δίδονται, δίνονται και σχετικές εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Στην πρακτική οι πληροφορίες αυτές δίδονται από κοινού με τους εμπειρογνώμονες από τα διάφορα Υπουργεία. Αυτές λοιπόν οι εξηγήσει στην Ελβετία είναι πολύ σημαντικές είναι εμπεδομένες, κυρίως και διότι επιβεβαιώνονται από την κυβέρνηση, η οποία κάθε φορά αποτελείται από πολλά και διαφορετικά κόμματα και κατόπιν τούτου μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι σε κάθε θέμα ε, ε υπάρχει μια αντικειμενικότητα, όλες οι τοπικές κυβερνήσεις ε, προφανώς ενδιαφέρονται και οι δικές τους εξηγήσεις να περιλαμβάνονται στις εξηγήσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ε, για την αποδοχή των εξηγήσεων αυτών είναι το γεγονός ότι οι επιτροπές που διοργανώνουν το ε, δημοψήφισμα ε, επιτρέπουν περιθώριο έτσι ώστε τα επιχειρήματα να αναφέρονται με απόλυτη ευχέρεια. Έρχομαι τώρα στο συμπέρασμα το οποίο εξάγω. Λόγω όλων αυτών λοιπόν προκύπτουν κατά τη δική μου άποψη τέσσερις συστάσεις ε, για τη δημιουργία της απαραίτητης ε, υποδομής έτσι ώστε να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάω λοιπόν με το θέμα της ε, ενημέρωσης. Για να υπάρχει μια ισόρροπη ενημέρωση πρέπει στις ψηφοφορίες, να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή και νομίζω ότι το παράδειγμα της Ελβετίας και του Bundesrat ε, στις ε, περισσότερες περιπτώσεις ε, είναι ένα παράδειγμα αποδεκτό και πιστεύω όπως και στην Ιρλανδία μπορεί να υπάρχει μια επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται της ε, ενημέρωσης. Μια τέτοια λοιπόν επιτροπή του δημοψηφίσματος ε, έχει ως υποχρέωση πρώτα να ε, προετοιμάσει το θέμα, να δημοσιευτεί ένα φυλάδιο ψηφοφορίας και επίσης καλείται η Επιτροπή αυτή να λαμβάνει υπόψη της και τα υπέρ και κατά επιχειρήματα. Η δεύτερη λειτουργία μιας τέτοιας Επιτροπής είναι να φροντίσει κανείς ε, για την ε, προσέλευση, για τη συμμετοχή, ε, να δίνονται πληροφορίες για το πώς ακριβώς πρέπει να γίνεται η ψηφοφορία, ποιος μπορεί να συμμετέχει και πώς ακριβώς μπορούν να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση και στις άμεσα ενδιαφερόμενες πληθυσμιακές ομάδες. Όσον αφορά τώρα τη σύνθεση της Επιτροπής, έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις. Η Επιτροπή μετά από εντολή του διαμεσολαβητή μπορεί να συγκληθεί από το ίδιο το Κοινοβούλιο και αποφασίζει ο ε, διαμεσολαβητής. Παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος μπορεί να είναι πρώην ε, δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η δεύτερη σύσταση που θέλω να καταθέσω είναι η εξής παράλληλα με τις ε, επιτροπές δημοψηφίσματος που συστήνονται ad hoc, είναι καλό να υπάρχει και μια συμβουλευτική επιτροπή και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο εφόσον ε, πρέπει ε, να υπάρχουν, θεωρείται κρίσιμο ότι πρέπει να υπάρχει μια ένας φορέας ο οποίος μπορεί ακριβώς να λαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία να παρακολουθεί τις επιτροπές των δημοψηφισμάτων. Ε, να γίνεται επίσημος έλεγχος ε, και επίσης και να υποστηρίζει την ε, μετάφραση των κειμένων. Στους πολίτες μια τέτοια, ένας τέτοιος φορέας πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης και πρέπει να είναι και αρκετά μετριοπαθής. Ποτέ δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι πρέπει να επηρεάζεται μια επιτροπή που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Επίσης, ένας τέτοιος φορέας πρέπει να είναι ή δυνατόν ανεξάρτητος, πολιτικά ανεξάρτητος ε, και ε, πρέπει να μην επηρεάζεται από εντολές. Νομίζω λοιπόν ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τέτοια επιτροπή ε, θα πρέπει να συσταθεί. Η τρίτη μου σύσταση είναι η εξής. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει εύρυθμη συνεργασία, ε, να υπάρχει ε, έλεγχος των υπογραφών. Γιατί ε, όταν πρόκειται για την άμεση δημοκρατία, εκείνο που παίζει ρόλο είναι κατά κύριο λόγο η νομολογία. Η νομολογία πρέπει να είναι και νομιμοποιημένη. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι διασφαλισμένο ότι σε αυτή την νομολογία θα συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου και να μην είναι ο ίδιος ο οποίος ε, θα συμμετέχει περισσότερες φορές στην ίδια διαδικασία και με τον τρόπο αυτό να αποκτά κάποιο πλεονέκτημα. Φτάνω στο τελευταίο σημείο της ε, παρατήρησής μου. Η εμπειρία δείχνει ότι τα δημοψηφίσματα ενέχουν, ε, περιλαμβάνουν ε, ένα τεράστιο πολιτικό δυναμικό. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι αν δει κανεί την πρακτική εκ του μακρόθεν, και εάν ασχολείται κανείς με μία επιτροπή η οποία διεξάγει δημοψηφίσματα, παρουσιάζονται περιπτώσεις χειραγώγησης, ε, παραδείγματος χάρη κατά τη διαδικασία ε, της καταμέτρησης ψήφων ε, τόσο σε νομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο πρέπει να ληφθούν μέτρα για τέτοιου, τέτοιες μορφής λαθροχειρίες. Εάν ασκείται η προσπάθεια άσκησης επιρροής, θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις. Από οργανωτικής πλευράς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι ε, υπογραφές ε, πρέπει να διασφαλίζονται και επίσης ε, και ο χώρος συλλογής των πληροφοριών θα πρέπει να είναι μυστικός. Συνοψίζοντας λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η δική μου σύσταση είναι να υπάρχει μια ad hoc επιτροπή δημοψηφισμάτων, η οποία θα είναι αρμόδια για την ενημέρωση να υπάρχει ένας, ε, μια μόνιμη συντονιστική υπηρεσία η οποία να είναι ουδέτερη. Επίσης ε, να υπάρχει μια αξιόπιστη υποδομή για να ελέγχονται υπογραφές και τέλος ε, να υπάρχουν νομικές προδιαγραφές που θα εξετάζουν το θέμα της πρωτοβουλίας να μπορούν να απορρίψουν οποιασδήποτε προσπάθειες χειραγώγησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Nagyon szépen köszönöm. Rendkívül értékes volt mind három Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικές και οι παρουσιάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, καθηγητές μας και να κηρύξω τώρα την έναρξη του γύρου των ερωταπαντήσεων. Πρώτα απ' όλα, θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου και ευρωβουλευτές εάν θέλουν να σχολιάσουν να ρωτήσουν κάτι. Κύριε Μπρόνς, φυσικά και έχετε το λόγο. Ναι, νομίζω ότι ε, ήταν ε, σχεδόν υποχρεωτικό να μιλήσω. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε διάλογο για αυτό το θέμα. Δεν ε, περιέγραψα εγώ... Δεν θα περιέγραφα την κίνηση των δημοψηφισμάτων από τις κυβερνήσεις ως δημοκρατική, άμεση δημοκρατία. Αντίθετα, αντιδημοκρατική τη διαδικασία θα την, θα τη θεωρούσα, Τέλος πάντων, υπήρξε ίσω μια παρανόηση πάνω σε αυτό. Άκουσα κάτι ενδιαφέρον από τον κύριο Γκρό. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η ελευθερία διαλόγου δεν εγγυάται την αλλαγή. Η απουσία όμως ελευθερίας, γιατί σε σχέση δηλαδή με τη διατύπωση ερωτήσεων, αποτρέπει την αλλαγή. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είπατε αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ασκεί κριτική ε, στην ε, μη ε, έγκριση κάποιων πρωτοβουλειών των πολιτών. Δηλαδή, αν υπάρχει εξουσία να αρνούνται για διάφορους λόγους τις πρωτοβουλίες των πολιτών, είτε γιατί δεν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίε, γιατί είναι δευτερεύουσε, είτε με βάση αυτά που λέει ο κ. Σεύκοβιτς, ότι είναι κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο ερώτημα προς, προς, προς την δόκτωρα Μπράουν Μπίντερ. Σε ό,τι αφορά τη συλλογή των 50.000 υπογραφών. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι οργανώτες θα προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν παραπάνω, γιατί κάποιες από αυτές μπορεί να ακυρωθούν. Άρα σίγουρα θα θέλουν να ε, συγκεντρώσουν μεγαλύτερο αριθμό. Υπάρχει ε, κάποιο στοιχείο για το ποσοστό των ε, υπογραφών που ακυρώνονται. Είναι 5% παραπάνω. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον Κέραντ Χέφνερ τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί εμπειρογνώμονες, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει σχέση με την εισήγηση η Και σας ε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, κυρία Λίμπε, για το γεγονός ότι... Έχουμε εδώ τους ε, πρωταγωνιστές της άμεσης δημοκρατίας και της ε, συμμετοχικής, αν θέλετε, το πούμε, δημοκρατίας που συλλογίζεται, που κάνει σκέψεις, ε, διότι θα πρέπει να δούμε όλη την εργαλειοθήκη αν θέλουμε να καταλήξουμε στο τι ακριβώς ε, θα σημάνουν αυτά στο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας ερωτήσω κατά πόσον εσείς μεταξύ σας ε, κάνετε κάποια ε, συγκεκριμένα βήματα ή μήπως ε, απλά είσαστε δογματικοί σε αυτό που πιστεύετε. Δηλαδή, να το πω με άλλα λόγια, η συμμετοχική δημοκρατία δεν νομίζω ότι αποκλεί του αντίον συνοδεύει όλα τα άλλα μέτρα. Η δική μου εμπειρία, η άμεση εμπειρία με την συμμετοχική αυτή δημοκρατία είναι η εξής. Εγώ ταχθηκα υπέρ της άμεσης δημοκρατίας στη Γερμανία. Τότε όμως δεν είχαμε ε, μεγάλη εμπειρία και είχα προσκληθεί ε, σε μία ε, συζήτηση τότε από μία εφημερίδα που δεν υπάρχει πια με έναν συνάδελφο ο οποίος ακριβώς όπως και εγώ έπαιζε τότε σημαντικό ρόλο στην, στο κίνημα της πρωτοβουλίας των πολιτών. Και ήταν μία πολύ έντονη διαμάχη γιατί είχαμε πει ότι και σκεφτεί έχουμε ε, πάρα πολλές ε, δραστηριότητες και τώρα έρχεται ο Χέφνερ και θέλει όλα αυτά να τα εντάξει μέσα σε ένα πλαίσιο και ξέρετε τι θα γίνει. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα καταπνιγούν διότι θα είμαστε αναγκασμένοι ε, να ακολουθούμε μία συγκεκριμένη γραμμή. Στην Αυστρία η, κατά το πρώτο δημοψήφισμα ε, τι ακριβώς ε, συνέβαινε και βοήθησα κι εγώ στον, ε, στη μάχη ε, πριν από την ψηφορία όταν επρόκειτο για την απόσυρση της Αυστρίας από πυρηνικά προγράμματα. Ξαφνικά λοιπόν προέκυψαν περισσότερες ε, κοινωνικές πρωτοβουλίες από ό,τι υπήρξαν ποτέ στην ιστορία της Αυστρίας. Παντού γινόντουσαν συζητήσεις, δημιουργούνται ομάδες, ε, δηλαδή ε, δεν μπορούσε κανείς ε, καν να βγει από το τρένο ε, χωρίς να πέσει πάνω σε κάποιον που να μοιράζει αν θέλετε φυλάδια. Η δική μου λοιπόν η εντύπωση είναι ότι Ποτέ δεν προκύπτουν τόσο πολλές συζητήσει ε, όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το τέλος θα προκύψει δημοψήφισμα έτσι και αλλιώ. Αυτά λοιπόν είναι δύο στοιχεία τα οποία ταιριάζουν και όπου το ένα θα μπορούσε να προετοιμάσει το άλλο. Το δεύτερο ερώτημα που έχω είναι το εξής ε, και αυτό ε, θα ήθελα να την υποβάλω στον Ανδρέας Γκρός και στην Άντια Μπχόμπιντα. Κυρία Μπίντα, ε, σε αυτή την, ε, σε σαφή αυτή τη διαδικασία και το βρίσκω ε, πάρα πολύ χρήσιμο ο αντικρό ε, έθιξε τα βασικά θέματα. Το δικό μου το ερώτημα είναι, αν βέβαια θέλετε να τοποθετηθείτε από αυτού, πώς, ε, πώς μπορεί να, ε, ποια μπορεί να είναι η έκβαση ενός ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος. Έχετε κατά νου την τάξη μεγέθους, το τι απαιτείται για να διοργανωθεί κάτι τέτοιο, το χρονικό διάστημα, ε, τα αποτέλεσμα, γιατί ένα ευρωπαϊκό ε, δημοψηφισμό είναι τελείως διαφορετικό από ένα εθνικό ε, ή σε επίπεδο καντονίου. Και κυρίως όταν πρόκειται για θέματα της συνθήκης, όπου το ερώτημα που θα τίθεται είναι και κατά πόσον όλα αυτά θα ισχύουν και στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε λιγάκι με τις προτάσεις σας. Ωραία. Κλείνει ο κύκλο αυτό. Έχω και εγώ βέβαια κάποιε ερωτήσει, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να δώσετε ήδη τις απαντήσεις σα στα πρώτα ερωτήματα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γιατί σε όλους απευθύνθηκαν τα ερωτήματα. Να αρχίσουμε από αριστερά προ τα δεξιά. Υπάρχει ένα ερώτημα για το κατά πόσον αυτοί που υποστηρίζουμε την άμεση δημοκρατία και αυτοί που υποστηρίζουν την διαβουλευτική δημοκρατία, αν μπορούμε να συνομιλήσουμε και αν υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη. Εγώ από τη δική μου σκοπιά θα έλεγα το εξή για την άμεση δημοκρατική διαδικασία. Για να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση χρειάζονται υποδομές. Διατάξεις που θα βελτιώνουν και θα προασπίζουν ε, την ασφάλεια της διαβούλευσης, το άνοιγμα της διαδικασίας, να είναι ανοιχτή δηλαδή ενώ η διαδικασία. Όποιοι θέλουν να μπορούν να έχουν λόγο, να είναι ισότιμο το πεδίο, να υπάρχει διαφάνεια, να παρέχεται ενημέρωση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, κύριε Γκρός, και είναι μάλλον πρόβλημα όταν μιλάω ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τα δημοψηφίσματα επικύρωσης Θέλουμε να παρεμβαίνει το κοινοβούλιο, αν δεν παρεμβαίνει το κατηγορούμενο, από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε ε, να κλέψει, αν θέλετε, αυτό την όλη διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν ε, κάποια δυσκολίε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, θα έλεγα και πιο επιτεδευμένους κανόνε για τη διάρθρωση τη δημόσια ενημέρωση και επικοινωνία σε μικρό ή πολύ μικρά ακροατήρια και βήματα συζήτησης. Τώρα, αν χρειάζεται να γίνονται δημοσίσματα ή όχι τελικά. Φυσικά μπορεί το δημοσίσμα να είναι ένα ισχυρό κίνητρο να συμμετάσχει ο κόσμος. Μπορεί επίσης όπως στη Στουτουκάρδη για, για το σταθμό, για το, για το σιδηρόδρομο Στουτουκάρδη 21, υπήρξε μεγάλη πόλωση στη, στη δεν ήταν υποχρεωτικό το δημοψήφισμα, ήταν προαιρετικό. Γιατί τον τελικό λόγο θα τον είχε περιφερειακή κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, Ο ρόλος αυτών των διαβουλευτικών μεθόδων είναι ευρύτερο το πεδίο. Είναι προϋπόθεση για τις δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά πηγαίνει πιο πέρα ακόμη και το διαβουλευτικό μήνυμα πρέπει να συμπεριληφθεί νομίζω και στη διαδικασία της αντιπροσώπευσης. Είναι κάτι το συνεχές στις διαδικασίες. Δηλαδή, Βέβαια έχουμε το Europe Direct, ε, κάτι που χρησιμοποιούμε για πολύ ζωντανέ ε, συζητήσεις, ε, παρουσία βουλευτών ήμελών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής και τοπικών προσώπων στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τοπικών ενδιαφερομένων φορέων. Άρα δεν δίνουμε μόνο περί ε, πληροφόρηση, είναι και ένα βήμα συζήτηση. Και καλό θα ήταν αυτό το εργαλείο να συνδεθεί και με τη λήψη αποφάσεων συγκεκριμένα. Γιατί κάποιε φορέ οι βουλευτέ το χρησιμοποιούν και ε, προσπαθούν έτσι να δοκιμάσουν, να κάνουν, ε, αν θέλετε, μια ανείχνευση του εδάφους. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Κύριος Γκρός. Να απαντήσω στον κύριο Μπρόν. Χαίρομαι πολύ καλά γιατί με καταλάβατε πολύ καλά κι εσείς. Ήθελα να δείξω ότι η εξουσία να επιβάλλει κανείς τη διεξαγωγή συζήτηση είναι μια τεράστια δύναμη. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι άμεσα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Και υποτιμούν τη συζήτηση, δεν καταλαβαίνουν την αυταξία της συζήτησης. Και θα έλεγα το εξή. Χωρί συζήτηση, χωρί διάλογο, αλλαγή δεν γίνεται. Ο διάλογο, η συζήτηση είναι εγγύηση αλλαγής. Είναι προαπαιτούμενο. Και για να μπορεί κανείς να επηρεάσει αυτό που ο απλός άνθρωπος στην κουζίνα του σπιτιού του, ε, στο σταθμό, στο λεωφορείο συζητά, είναι τεράστιο. Είναι τεράστια δύναμη. Και ξέρω ότι υπάρχει μετά εκθετική ε, αύξηση του όγκου αυτής της συζήτησης. Και αυτό είναι και το επίκεντρο της όλης συζήτησης. Και το δεύτερο είναι το εξής. Όταν κανείς προσπαθεί να καταλάβει τι θα πει δικαιοσύνη. Είπατε ότι ε, κάποια πράγματα και το πρωί, κύριε Χέφνερ. Πόσοι και πόσοι δεν ε, καταγγέλνουν, δεν ακούγονται, δεν ακούγεται, δεν ακούγεται η φωνή τους. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο να λέει κανείς κάτι, αλλά και να μπορεί να το ακούσει κάποιος άλλος αυτό που λέει. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο κρίσιμα προβλήματα. Και αυτό ε, το καταγγέλνουν οι περισσότεροι. Όταν του ρωτά κανεί γιατί είστε εξοργισμένοι, αυτό καταγγέλνουν, ότι δεν του ακούνε. Δεν ακούγεται τη φωνή του. Και νομίζω ότι αυτό είναι στην καρδιά του όλου ζητήματο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Για να ακούγεται τη φωνή μα. Και δεν είναι τελευταία αυτά. Δεν είναι κάτι σύγχρονο. Είδα το 19ο αιώνα. Τα έλεγαν στην Ελβετία και στη ΣΥΠΑ αυτοί οι οποίοι κατέκτησαν τα δικαιώματα αυτά για ολόκληρο το λαό. Λέγεται πολλέ φορέ τα ζητήματα που αφορούν το λαό είναι τόσο σημαντικά που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στο λαό. Και οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί είναι στην ίδια μονάδα του νοσοκομείου. Πάσχουν από το ίδιο νόσημα, θα έλεγα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το ερώτημα ε, των, ε, του στοχασμού και των συζητήσεων, θέλω να πω ότι ε, υπάρχει μία αντίφαση ανάμεσα στις συζητήσεις και στην άμεση δημοκρατία, διότι η επικοινωνιακή δύναμη είναι το καθοριστικό στοιχείο της ε, άμεσης δημοκρατίας. Ε, στην θεωρία της ε, συμμετοχικής, ας την πούμε, δημοκρατίας, deliberative είναι στα αγγλικά, αναφέρεται ότι πρόκειται για μία διεργασία που αφορά πολλά εκατομμύρια ή υπάρχουν εκείνοι που συρρυκνώνουν αυτό σε ένα και μόνο κομμάτι του πληθυσμού, σε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο κομμάτι αυτό οργανώνει τις ε, συζητήσεις. Και αν αυτό ε, το αμφισβητήσει κανείς, πρόκειται για μια ειδική μορφή της εκπροσώπησης ε, ή ξεκινάει κανείς με, μια, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, αμοιβόμενο, και αυτό όμως γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και εμείς μιλάμε για συμμετοχική δημοκρατία με την έννοια της ε, ε, διάδοσης. Ο Τόνι Μπλερ το εκμεταλλεύτηκε αυτό χρόνια ολόκληρα, όπου κάθε ιδέα πριν έρθει στο κοινοβούλιο τη δοκίμαζε σε τέτοιου είδους ομάδες. Και αυτό δεν απελευθερώνει, Αυτά, απλά αυτό είναι μια ε, εκμετάλλευση τελειοθυρίας των κυβερνήσεων. Έτσι λοιπόν αυτό το δεύτερο επίπεδο της εκπροσώπησης δεν πρέπει κανείς να το πουλάει ως εκδημοκρατισμό γιατί εμείς επιθυμούμε όλοι οι άνθρωποι και όχι κάποιοι αιρετοί να είναι ελεύθεροι και να μην είναι ελεύθεροι στη θέση κάποιων άλλων. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Αλλά και εγώ συμφωνώ ότι τις σύγχρονες τεχνολογίες ε, πρέπει κανείς ε, να τις συμπεριλάβει ως συμβολή και όχι ως υποκατάστατο. Αυτή η συζήτηση ε, έχει γίνει στη Γερμανία πριν από 15-20 χρόνια, ε, πριν εμφανιστεί η λέξη deliberation. Ο Ντίντλ στη Γερμανία το ανέφερε αυτό και ήθελε να το πουλήσει ως υποκατάστατο της ε, δημοκρατίας. Δεν είναι υποκατάστατο, συμπλήρωμα θα μπορούσε να είναι. Τώρα, τα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα ε, μπορείτε να δώσετε εντολή, ε, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν στοιχεία που πρέπει κανείς να τα προσέξει πάρα πολύ. Παραδείγματο χάρη, δεν πρέπει να μαζεύονται πάρα πολλές υπογραφές. Όμως ε, οι υπογραφές πρέπει να μαζεύονται από διάφορες χώρες. Ακόμα και αν αυτό είναι επίπονο, αυτό είναι μια προϋπόθεση που προάγει ε, το ευρωπαϊκό και περιορίζει το εθνικιστικό και επίσης ε, θα πρέπει κανείς να απευθύνεται και σε μικρές ομάδες, όχι μόνο σε μεγάλες, δηλαδή σε συνδικάτα, στο ΒΒΕΦ και σε άλλους. Ε, ε όχι ένα 10 ή 20% για να γίνει όμως αυτό, είναι χρονοβόρη διαδικασία, πενταετής αν θέλετε. Κυρίως στην Ευρώπη όπου ακόμα δεν υπάρχει τέτοιος ε, πολιτισμός ε, και για το Κοινοβούλιο, για τις αρχές, ε, για τις κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρχει πάντα χρόνος. Στα 15 αυτά λεπτά στα 15 αυτά λεπτά δεν μπορέσαμε να καταδείξουμε τι ακριβώς συμβαίνει το ίμιση ε, των δημοψηφισμάτων στην Ελβετία είναι αποτελεσματικά και όσο πιο γρήγορα όμως ε, γίνεται κάτι, τόσο μικρότερο το αποτέλεσμα. Αν θέλει πραγματικά κανείς να ασκήσει επιρροή, ε, πρέπει να έρθει σε αντιπαράθεση κανείς με το αντικείμενο. Αυτό είναι το αντίθετο με την πραγματικότητα της ε, Καλιφόρνιας, όπου μπορεί κανείς να καταθέσει μία πρόταση το Μάρτιο και μετά να ψηφίζει ήδη το Νοέμβριο και δεν γίνεται τίποτα πέρα από μία μεγάλη μάχη στην τηλεόραση. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την πλειοψηφία, θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση όσον αφορά το συνταγματικό επίπεδο με το επίπεδο του νόμου. Το επίπεδο του νόμου και εκεί ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει μία πλειοψηφία ε, όταν όμως πρόκειται για το Σύνταγμα και θέλω να κάνω εδώ μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε Σύνταγμα και σε ένα είδος ε, συνταγματικού συμβολέου. Όταν πρόκειται για το πραγματικό Σύνταγμα θα πρέπει να είναι ε, σαφές ότι πρέπει να έχουν ε, συνενέσει οι πολίτες ε, ένα κείμενο αν θέλετε 400 σελίδων που ε, κανείς δεν το έχει διαβάσει. Στην Δανία όμως δεν είχαν το κείμενο και επειδή ήταν και ακατανόητο ψήφισαν όχι. Στην Αλβετία, αν δεν είναι διατυπωμένο σωστά το κείμενο, είναι πολύ πιθανόν όλοι να ψηφίσουν όχι τα, οι νόμοι πρέπει να είναι κατανοητοί και αυτό συμβαίνει σε εμά. Όχι επειδή είμαστε καλοί στην έκφραση, κάθε άλλο, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι αν δεν έχουμε σαφή ε, επεξήγηση των νόμων, ε, δεν μπορούμε και να πείσουμε τους νόμους να υπερψηφίσουν. Επίσης, ε, είναι σαφές ότι όσον αφορά τις ε, συνθήκες ή το σύνταγμα αυτό καθ' αυτό, προφανώς και πρέπει να υπάρχει μια δημοκρατική εξέλιξη. Και τίθεται και το εξής ε, ερώτημα. Η Ελβετία έχει τις ε, δικές της δυνατότητες να τα ελέγξει όλα αυτά. Θα πρέπει βεβαίως να είμαστε ισότιμοι με την Μάλτα και με τη Γερμανία, αλλά παρόλα αυτά αν θέλετε είναι μια ευνοϊκή θέση των μικρών. Και αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουν οι μεγάλοι ποσοτικά για να ενσωματωθούν όλοι. Και στην ε, Ελβετία, η Ζηρίχη, ας πούμε, έχει 1,1 εκατομμύριο κατοίκους και αυτοί έχουν τον ίδιο ψήφο, το, την ίδια δύναμη όπως ένα άλλο καντόνι που έχει μόνο 30.000, αν θέλετε. Ε, διότι αν δεν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε στο ίδιο επίπεδο τα μικρά κράτη με τα μεγάλα. Ε, υπάρχει αλλιώς ο κίνδυνος τα μικρά κράτη να φοβούνται ότι θα τα καπελώσουν τα μεγάλα σε όγκο. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ σύντομα ε, σε αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως ε, για τα ποσοστά και για τις ε, υπογραφές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι υπάρχει έλεγχο σε δύο επίπεδα. Ε, το πρώτο επίπεδο είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση και ο δεύτερο έλεγχο είναι σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το ομοσπονδιακό επίπεδο ελέγχει κατά πόσον ο Δήμο η κοινότητα έκανε καλά τη δουλειά τη και μήπω υπάρχουν προβλήματα. Ε, όσον αφορά τον δεύτερο έλεγχο, εδώ κατά κανόνα δεν προκύπτουν άκυρες ε, ψήφοι. Ε, κάτω από 1% αν θέλετε. Στο πρώτο επίπεδο το αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον οι επιτροπές ανάληψης πρωτοβουλίας έχουν κάνει σοβαρά τη δουλειά τους, ε, κατά πόσον έχουν ψηφίσει σωστά. Να μην ας πούμε ψηφίζει κάποιος Donald Duck, αυτό δεν είναι έγκυρη ψήφος. Και εκεί λοιπόν ε, κατά κανόνα οι Επιτροπή επιτροπές ε, δημοψηφίσματος ε, κάνουν ε, πολύ καλή δουλειά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων. Όσον αφορά, μάλλον, να πω και άλλες δύο σκέψεις που είναι συμπληρωματικέ σε αυτά που ελέγχθησαν μέχρι τώρα σχετικά με τα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα και την αποκαλούμενη συμμετοχική δημοκρατία. Όσον αφορά λοιπόν την διαβουλευτική οικονομία, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε, ε, να προβούμε στη συγκέντρωση ε, ψήφων και η εμπειρία έχει καταδείξει ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει κανείς ε, ψήφους. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατά την άποψή μου στην ε, συμμετοχική διαβουλευτική δημοκρατία υπάρχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας. Και επειδή υπάρχει αυτό, επιβάλλει κανείς ε, ήδη εκ των προτέρων την αντιπαράθεση με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Γιατί δεν θέλει κανείς να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Άρα δηλαδή τι σημαίνει ότι συζητά εκ των προτέρων με τους ε, πολίτες. Δεύτερη σκέψη. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα όσον αφορά ε, στο δικαίωμα κατάθεσης ε, πρότασης, να προτείνει κανείς ένα συνταγματικό ε, δικαίωμα. Νομίζω ότι δεν κερδίζει κανείς τίποτα αν προβλέψει την προθεσμία των έξι μηνών. Αυτό απλά δυσκολεύει ε, τα πράγματα και δεν διευκολύνει ούτε την κατανόηση ούτε την υποστήριξη. 18 ε, μήνες έχει κανείς ε, χρόνο στην Ελβετία για κάτω από χίλιες ψήφους και ήδη αυτό είναι πρόβλημα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι όσον αφορά αυτό το τελευταίο παράδειγμα, έχουμε την European Citizens Initiative ε, και μπορούμε να δούμε ε, πόσο γρήγορα ε, μπορεί κανείς να προχωρήσει με τις ηλεκτρονικές, ηλεκτρονική υπογραφή. szeretnék kérdést feltenni. E, Υπήρχε μια ερώτηση προς τον κύριο Γκρός, ε, την οποία θέλω να θέσω. Η άμεση δημοκρατία δεν είναι αναλλακτική της, συμπληρωμα... της δημοκρατίας, αλλά είναι συμπληρωματικές έννοιες, αλληλοενισχύονται όπως είπατε. Το Γερμανικό Σταγματικό Δικαστήριο, στην απόφαση του για τη Λισαβόνα, επισημαίνει την ανάγκη αντιπροσωπευτικότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η απόφαση ισχύει και για ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή η νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού ε, ε, Κοινοβουλίου θα αυξηθεί με την άμεση δημοκρατία. Πολύπλοκο είναι το ερώτημα, αλλά υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα. Επίσης είπατε ότι είναι σε κρίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και η δημοκρατία σε κρίση τελικά. κατά τη δική σας την κρίση. Πρόκειται για κρίση της δημοκρατίας, αυτής καθεαυτής. Ο πρώτος ομιλητής, ε, συγκεκριμένα η ε, πρώτη ομιλήτρια, έκανε το εξής ερώτημα. Τι έχει μείνει ε, από τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Είπε για έναν ολοκλήρωτο ταξίδι, ένα ταξίδι που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Υπάρχουν απτές προτάσεις. Ποιες πρέπει να προωθήσουμε ως χαράκτης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διορθώσουμε τα πράγματα και βελτιώσουμε την κατάσταση που εσείς μας σχεδι... Ε, σκιαγραφίσατε. Πολλά είναι τα επιχείρηματα που αναφέρατε. Μεταξύ αυτών μιλήσατε για την ευθύνη, τη λογοδοσία. Και είπατε ότι είναι ένα πάρα πολύ ε, έντονο αίτημα και θεμητή διεκδίκηση από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος Γκρόση είπε ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο οι εκλογές. Είναι κάτι παραπάνω, γιατί μας επιτρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Καταλαβαίνει όμως ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ελευθερία αυτή. Γιατί πρόσφατα είχαμε πολλές εξελίξεις. Και πραγματικά εγώ βάζω ένα ερωτηματικό στο κατά πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται τελικά το τι είναι στη δημοκρατία. Ιδίω οι νέοι που δεν έχουν ζήσει τον πόλεμο, οι νέε γενιέ δεν έχουν ζήσει πόλεμο και εννοούν διαφορετικά, καταλαβαίνουν διαφορετικά τη δημοκρατία από όσους έχουν βιώσει πολέμους. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω. Και δεν απευθυνόμαστε στον κύριο Γκρός, αλλά και στις δύο κυρίες. Ευχαριστώ. I'm very grateful for these questions because... Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, ερωτήσεις, γιατί μπαίνουν πραγματικά στην ουσία της ε, συζήτησης. Μαζί με τον φίλο και συνάδελφο τον κύριο Σίλε συζητήσαμε κάθε απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και συμφωνήσαμε πως είναι ένα από αυτά τα δικαστήρια που ποτέ δεν ε, θα έφερνε αντίρρηση στη δημιουργία μιας δημοκρατικής πολιτείας σε υπερεθνικό επίπεδο. Η αντίρρησή τους είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χέφνερ στις παρατηρήσεις του. Όταν υπερεθνικοποιούνται όλο και περισσότερες πολιτικές χωρίς να υπάρχει ένα δημοκρατικό βάθρο τότε υπάρχει η αντίθεση του δικαστηρίου αλλά όταν υπάρχει και δημοκρατία στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργείται ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα και όπως είπα η άμεση δημοκρατία θα κάνει οποιαδήποτε αντιπροσώπευση πιο αντιπροσωπευτική, γιατί το ξέρει και η κυρία Μπράουν, στην Ελβετία πρέπει κάθε βράδυ να συζητάμε ε, τρεις μήνες πριν ε, ψηφίσουμε οτιδήποτε. Πάμε και συζητάμε με τους πολίτες, γιατί ξέρουν πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την στήριξη των πολιτών. Είναι τελείως διαφορετική η σχέση και πολύ μικρότερη η απόσταση με το να συζητάμε ένα ζήτημα. Ακούμε όλα τα άλλα πράγματα που ανησυχούν τους πολίτες. Υπ' αυτή την έννοια ένας βουλευτής ξέρει το τι θέλουν από αυτόν οι, άνθρωποι και μπορεί βεβαίως να κινηθεί αναλόγως. Και υπ' αυτή την έννοια το, το γερμανικό δικαστήριο α, είμαι σίγουρος πως δεν θα είχε αντίρρηση. Γιατί αντιλαμβάνεται και το πώς μπορεί να διαμεριστεί η εξουσία μεταξύ διαφορετικών επίπεδων. Γιατί έχουν μια ομοσπονδιακή παιδεία ε, ε, αφού είναι Γερμανοί. Επίσης για τέταρτη φορά υπέβαλα μία έκθεση για την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ευρώπη στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία αλλά και η δημοκρατία χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό αν όχι ένα παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί όπως είπα η υπόσχεση ουσιαστική για τις ευκαιρίες Τη δημοκρατία δεν μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα στο εθνικό επίπεδο, γιατί η οικονομία είναι διεθνή. Μπορεί να είναι τοπική η πολιτική, αλλά η οικονομία είναι διεθνή. Ήδη πριν από 20 χρόνια ο δήμαρχος του Αμβούργου είχε πει πως η εθνική δημοκρατία σήμερα είναι σαν να λέμε πως ε, είναι, έφερε ένα παράδειγμα, πως η Εθνική Δημοκρατία είναι πλέον σαν το πιδάλιο ενό πλοίου που είναι έξω από το νερό. Δεν μπορεί πλέον να στρίψει το πλοίο. Οπότε κάποιοι λένε πως δεν μας χρειάζεται το πιδάλιο. Όχι. Εμείς θέλουμε πρέπει να φτάσει το πιδάλιο μέσα στο νερό, να επιμηκυνθεί. Γιατί ε, ξεκίνησε βεβαίως πριν από κάποιους αιώνες στη... στις Ιταλικές πόλεις η έννοια του, του κράτους, αλλά δεν λέει κανείς πως ε, το κράτος έθνος είναι το, το τέλος της δημοκρατίας. Και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω τη λέξη κρίση, γιατί μπορεί κανείς να πει πως σύγχρονες δημοκρατίες πάντα σε κρίση ήταν και το ίδιο μπορεί να πει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βρήκαμε πρόσφατα ένα άρθρο που είχε γραφτεί πριν από 25 χρόνια και μιλούσε για την κρίση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κάποιοι θα πούν πως ο μοντερνισμός είναι μία συνεχής κρίση, αλλά αν σκεφτόμαστε προσεκτικά τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη κρίση, είναι η ανεπάρκεια της μορφής και της ουσίας ο σημερινός κόσμος χρειάζεται μια άλλη πολιτεία, μια άλλη μορφή για να πραγματοποιήσει τις ελπίδες του κόσμου που εννοούμε με τη λέξη δημοκρατία. Γι' αυτό το εθνικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δεν επαρκούν πλέον. Και ίσως από αυτή την έννοια πρέπει να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε πιο ακριβείς όρους από τη λέξη κρίση, γιατί ναι, και η κρίση ισχύει, ισχύει βεβαίως. Γιατί εάν δεν υπάρχει ένα δημοκρατικό θεμέλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δεν θα έχει την απαραίτητη εξουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα θα επιλέγει ο κόσμο στο εθνικό κράτο. Γιατί θεωρεί πω εκεί πέρα θα βρει τη λύση. Παρά το ότι, όπω είπα, δεν ισχύει αυτό. Ένα τρίτο στοιχείο. Πρώτα απ' όλα, ως κάποιο, ο οποίος εργάζεται 17 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εντάξει, ίσως να μην γνωρίζουμε ένα τον άλλο τόσο καλά παρά το ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια όπω λέμε, νομίζω πω Ευρω... οι δυτικοευρωπαίοι υποτεμούν την κληρονομιά του ολοκληρωτισμού. Και υπ' αυτή την έννοια μπορεί να έχετε δίκιο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν διαφορετική αντίληψη της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αλλά από την άλλη, αν διαβάσει κανεί αυτά τα οποία έγραψε η Χάνα Άρεντ, ε, ενθαρρύνεται βεβαίως, γιατί αυτή βρήκε πολύ ελευθερία μετά την Ουγγρική επανάσταση μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αν παρατηρήσει κανείς τους ανθρώπους βλέπει πως ενστικτοδός έχουν μια υγιή αντίληψη της δημοκρατίας αλλά όταν ακούνε πάρα πολύ κάποιους πολιτικούς έχουν πρόβλημα να αντιληφθούν το τι σημαίνει και σήμερα ο δημόσιος λόγος έχει απαξιώσει κάπως αυτούς τους όρους ο κόσμος έχει πρόβλημα να, να καταλάβει αλλά νομίζω πως όταν έχει την ευκαιρία κανείς να συζητήσει με τον κόσμο έχει την ικανότητα να βρει μια κοινή γλώσσα συνεννόησης που είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτή από αυτή τη φθαρμένη έννοια του, της δημοκρατίας και του εθνικισμού που ακούει από πολλούς πολιτικούς. Σας ευχαριστώ. Ja, ich würde gerne äh, äh, auch noch Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, Εγώ είμαι φίλος, απόλυτος φίλος της ε, διαδικασίας ε, διαβουλεύσεων και αυτό το χρειαζόμαστε πηγόντως στην πολιτική. Αυτό εξάλλου είναι κάτι που δημιουργεί μηχανία στους ανθρώπους και εμένα παρεπιπτόντως. Και για μένα τα, το 1 τέταρτο της ζωής μου το έχω περάσει σε κοινοβούλια. Και το κοινοβούλιο που έρχεται από τη λέξη παρλάρε, μιλάω, όπου υποτίθεται ότι γίνονται συζητήσεις και μέσω αυτών αναζητά κανείς ε, την καλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε σε κοινοβούλια που δεν επιτρέπουν τον ανοιχτό διάλογο. Όσοι ε, παρακολουθούν τις συζητήσεις, ε, σωστά πιστεύουν ότι οι αποφάσεις έτσι και έχουν ληφθεί. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις των Επιτροπών ε, μέσω ε, του webstream. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτή την διαβουλευτική διαδικασία, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι την διαβούλευση να, το, να αντιμετωπίζουμε ως ένα ευρύτερο εργαλείο. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας υποβάλω ένα ερώτημα, διότι έχω ζήσει πολλά και θετικά παραδείγματα, αλλά και άλλα λιγότερο. Και θα σας ε, θα αναφερθώ σε ένα κίνδυνο που για μένα είναι ο μεγαλύτερος. Δηλαδή υπάρχει το ερώτημα τι είναι εκείνο που μας ε, προστατεύει σε τελική ανάλυση ε, την διαδικασία διαβουλεύσεων να την αντιμετωπίζουμε ως ένα είδος πλασίμπο. Και θα αναφερθώ στο παράδειγμα μιας ε, κυρίας, την της οποίας κάνετε γνωρίζω το όνομα, και πρόσφατα ήμασταν μαζί στο τρένο, ε, ήρθε και μου είπε, στο κύριο κύριος σα σας ξέρω από τηλεόραση και μου λέει, πρέπει να σας πω κάτι. Μου είπε λοιπόν ότι προέρχεται ή έχει προσκληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο ε, διανυκτερεύσεις σε τρεις ημέρες σε πρώτη τάξη ξενοδοχείο με εκατοντάδες πολιτών, οι οποίοι πρόκειτο να ερωτήσουν τι θέλουν να αλλάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα τα έγραφαν σε ένα πίνακα και θα τελείωνε η όλη συγκέντρωση και μετά από έξι μήνες ε, έγραψε αυτή μια επιστολή. Ε, τι έγινε τελικά με την ιστορία και κατέληγε η κυρία στο ότι τίποτα. Όλα αυτά ήταν ε, για το Θεαθήνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτές τις πράξεις μας δημιουργούμε αυτή την εντύπωση για την πολιτική, ότι είναι για το Θεαθήνε. Η κυρία αυτή που σας είπα έζησε αυτή την εμπειρία και προκαλούμε λοιπόν ε, προσδοκίες από την πολιτική γιατί κάποιος που έχει συμμετάσχει σε μια διαβουλευτική διαδικασία ε, προσδοκά ότι αυτά τα οποία είπε θα ληφθούν υπόψη στην ε, λήψη των αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν έχω το εξής ερώτημα. Ποια είναι τα κριτήρια ή αν θέλετε οι προϋποθέσεις που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την απογοήτευση και να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία και πώς μπορεί κανείς να συνδέσει τις ε, διαβουλευτικές διαδικασίες με διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων σε κοινοβούλια ή οπουδήποτε σήμερα λαμβάνονται οι δημοκρατικές ε, αποφάσεις, όπου υπάρχει δημοκρατική εξουσία. Το άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω και πάλι ε, θα ήθελα να το υποβάλω και στους δύο ομιλητές, τη Νάντια Μπρόμπιντα και στον Ανδρέας Γκρός. Εχθές. Ήμασταν σε αυτήν εδώ την Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων και συζητήσαμε για την πολυεπίπεδη ε, διακυβέρνηση για τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Μιλήσαμε επίσης για την τραπεζική, την φορολογική, την πολιτική ένωση. Όλη λοιπόν αυτή η διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι μια διαδικασία όπου οι πολίτες είναι απλοί θεατές. Οι ε, πολίτες δεν ερωτώνται, οι θεσμοί λαμβάνουν τις αποφάσεις και ρώτησα χτες το βράδυ τι θα γίνει με την συντακτική συνέλευση, με τη διαδικασία εκείνη όπου οι πολίτες μπορούν να συμπεριληφθούν στην όλη διαδικασία, όπου προβλέπεται χρόνος για διαβουλεύσεις, για όλα αυτά που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, για περισσότερη δημοκρατία, για να υπάρχουν ε, θεσμοί, ε, όλα τα απαραίτητα. Και χωρίς να θέλω να κατονομάζω συναδέλφου, η απάντηση ήταν ότι πράγματι η συντακτική συνέλευση ήταν μια πολύ καλή ιδέα, αλλά όχι τώρα. Δεν τη χρειαζόμαστε τώρα, δεν πρέπει να υπάρξει τώρα, διότι ε, κάτι τέτοιο θα είχε απρόβλεπτα αποτελέσματα και τώρα καλούμεθα να ξεπεράσουμε την κρίση, να ε, έχουμε πιο ασφαλή πιο ασφαλείς καταστάσεις και όταν τα έχουμε ξεπεράσει την κρίση, τότε πια θα μπορούμε να ε, οργανώσουμε συντακτική συνέλευση, διαβουλεύσεις, ε, συζητήσεις ή οι πολίτες να λαμβάνουν δημοκρατικές αποφάσεις, αλλά όχι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν το δικό μου το ερώτημα που θέτω είναι το εξής Μήπως θα έπρεπε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μήπως ε, τώρα ακριβώς θα έπρεπε να έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και που ανοίγουν τη συζήτηση έτσι ώστε να μην έχουμε μια πραγματική ουσιαστική συζήτηση και όχι ένα μονόδρομο στα αποτελέσματα. Μια διαδικασία λοιπόν η οποία θα επιτρέπει τη νομιμοποίηση μέσα από τη συζήτηση και μέσα από δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή είναι η ερώτηση που είχα να κάνω και άλλη μία η οποία είναι η εξής. Πώς μπορούμε μέσα από άμεση διαβουλευτική συμμετοχική διαδικασία να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Με την έννοια να ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ε, και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Πολλοί συνάδελφοι, πολλοί εξ αυτών που επιθυμούν η Ευρώπη να μην αποτύχει, αλλά η Ευρώπη να στεφτεί από επιτυχία, πολλοί από αυτούς φοβούνται τα δημοψηφίσματα, διότι φοβούνται ότι τα δημοψηφίσματα αυτά θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν και όχι μόνο αυτό, να οδηγήσουν σε κατάρρευση το ε, ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ιρλανδία, Γαλλία, παραδείγματο χάρη. Και γι' αυτό λοιπόν ε, θέτω το ερώτημα αντίστροφα. Μήπως ή αλλιώς, να το πω αλλιώς, καλύτερα να το πω στα γερμανικά. Πώς ε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε να δρομολογήσουμε μία διαδικασία έτσι ώστε μέσα από την ίδια τη διαδικασία να προκληθεί μεγαλύτερη διάθεση για την Ευρώπη, να προκύψουν συνένεση, και διάθεση για μια κοινή Ευρώπη. Ποιο θα έπρεπε να είναι το περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Ε, και τελειώνω με μια ερώτηση προς τον κύριο Ανδρέας Γκρός, γιατί ξέρω ότι εσύ έχεις τοποθετηθεί επανειλημμένα στο ερώτημα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Το όλο εγχείρημα αυτό περί Ευρωπαϊκού Συντάγματος ε, δεν έχει κλείσει, απλά έχει ε, ανασταλεί. Εγώ ερωτώ λοιπόν, μήπως πρέπει να το ξεχάσουμε ή μήπως πρέπει να το φέρουμε πάλι στο προσκήνιο. Και αν ναι, μια τέτοια διαδικασία, τι μορφή θα μπορούσε να λάβει. Θα... Ήθελα να ε, σας δώσω το λόγο. Ε, για να τα πω έτσι σύντομα, μας ε, λέτε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή, άμεση ε, δημοκρατία και διαβούλευση οδηγεί και στη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου. Θα σας πω τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η δημοκρατία, η κρίση της δημοκρατίας πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μιλάω για κρίση ε, με την αντικειμενική έννοια του όρου, αλλά και με την υποκειμενική ε, ε, έννοια του όρου. Υποκειμενικά γιατί δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα δεν είναι αυτά που λαμβάνουν τι αποφάσεις που θα έπρεπε να λαμβάνουν. Υπάρχει εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ανάθεση αρμοδιοτήτων. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο χάσμα. Υποκειμενικά βλέπουμε επίσης την απογοήτευση που και εσείς είπατε ότι υπάρχει απογοήτευση, αποστασιοποίηση των πολιτών και όχι μόνο ή κατά κύριο λόγο μόνο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως εκδηλώνεται με την αποχή σε ευρωεκλογέ, αλλά γενικά χαμηλή προσέλευση και σε εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογέ βέβαια. Μειωμένη εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Βέβαια υπάρχουν διακυμάνσεις και διαφορές σε κάποια ε, κράτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δημοφιλέστερο από την Εθνική Βουλή, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ανάτι την κρίση ε, και επειδή είπα για το τι έχει απομείνει από την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, εννοούσα όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα αυτό το ζήτημα και θα πει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε, να διαβολευτούμε για το τι σημαίνει δημοκρατία, υπό τις ε, σημερινές ε, ευρωπαϊκές συνθήκες και έχουμε διαφορετικές έννοιες. Δεν μιλάμε μόνο για ε, την άμεση, αντιπροσωπευτική, διαβολευτική δημοκρατία, αλλά μιλάμε και για την επιρεθνική δημοκρατία, την ομοσπονδιοποίηση, τον φοντεραλισμό. Μιλάμε για τις εθνικές δημοκρατίες, μιλάμε για τη διεθνή κοσμοπολιτική δημοκρατία κτλ. Πρέπει λοιπόν να γίνει δημόσια συζήτηση για το τι εστί δημοκρατία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η τρέχουσα κρίση, η χρηματοπιστωτική, οικονομική, η τραπεζική κρίση συγκαλύπτεται αν θέλετε κατά τρόπο κατά κάποιο τρόπο με μια συζήτηση που γίνεται για το δημοκρατικό έλλειμμα. Ήμουν σε ένα συνέδριο που διοργάνωσε η Deutsche Bank ε, στη Φραγκφούρτη και το ερώτημα ήταν ποιος ε, κυβερνά ε, τη Γερμανία. Η Ευρώπη, η γερμανική κυβέρνηση, το συνταγματικό δικαστήριο, μη ερετά, μη εκλεγμένα όργανα για πίσω από κλειστέ πόρτε. Ποιο τελικά κυβερνάει τη Γερμανία. Υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη αντιπαράθεση και σύγκρουση για το πώς θα μπορέσουμε να δαμάσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. πρέπει να βρούμε πού συμφωνούμε, που θέλουμε, πού περισσότερη ρύθμιση ή θεωρούμε ότι μήπως είναι πρόβλημα, ε, μέρος του προβλήματος η θεωρουμε οτι μηπως ειναι προβλημα μερος του προβληματος η ρυθμιση και όχι μέρος της λύσης. Πώς θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τα θέματα και πώς θα βρούμε δημοκρατικέ διαδικασίες για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε ειρηνικά, ε, χωρίς οικονομικούς νομισματικούς πολέμους, τα προβλήματα. Τελευταίο ερώτημα που μου απευθύνονται ήταν πώς η διαβούλευση σχετίζεται ή μπορεί να σχετιστεί με τη λήψη αποφάσεων. Τη δημοκρατική και την αντιπροσωπευτική και τη συμματοχική. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα υπερπίδησης μια λανθασμένης θα έλεγα παράθεσης της ε, νομιμοποίησης της δικαδικασίας με, τη νομιμοποίηση του αποτελέσματος. Input-output legitimacy. Τα βάζουμε μαζί αυτά τα δύο. Ένα μετά το άλλο. Πρέπει να αλλάξουμε αντιμετώπιση και νοοτροπία. Θα πρέπει να αλλάξουμε και την ε, ε αντίληψή μας για αυτή την έννοια ώστε και τα μη εκλεγμένα όργανα να μπορούν και να πρέπει βέβαια να λογοδοτούν στη δημόσια κοινή γνώμη μέσω διαβουλευτικών διαδικασιών. Για μέσα δημοκρατία δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό. Για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα που δεν ε, έχουν εκλεγεί. Λέω, ρωτάω, δεν ξέρω. Ε, και εδώ θα ολοκληρώσω. Um, thank uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θέλει να σχολιάσει να ρωτήσει κάτι ο συνάδελφος Μπρόνς. Παρακαλώ κύριε Μπρόνς. No, that was just a microphone. Όχι, όχι, το, το μικρόφωνο ήταν αυτό. Έχετε το λόγο. Αναρωτιέμαι αν συμφωνεί το πάνελ και αυτό αφορά βεβαίως την ε, διαβουλευτική δημοκρατία αν συμφωνεί πως η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς πλήρη ελευθερία επικοινωνίας. Δηλαδή να μην υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, ε, πέραν βεβαίως από την ενθάρρυνση της βίας. Όμως πρέπει να υπάρχει και ελευθερία να ακούει και να διαβάζει κανείς τα όσα λέγονται, κατά το οποίο βεβαίως υπονοεί ελευθερία πρόσβασης στα ΜΜΕ και το καθήκον να μεταδίδονται, ειδικά σε προεκλογική περίοδο, το τι λένε όλοι οι συμμετέχοντες. Θυμάμαι όταν δίδασκα εγώ πάντα θεωρούσα πως ο στόχος του καλού μαθήματος ήταν αν είχα μάθει εγώ κάτι που δίδασκα και ένας μαθητής μου είπε η ελευθερία του λόγου δεν είναι το δικαίωμά τους να λένε ό,τι θέλουν είναι το δικαίωμά μου να ακούω ό,τι έχουν πει και νομίζω πως είχε δίκιο αυτή η ελευθερία πρέπει να υποστηριχθεί ευχαριστώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπρόνς. Άλλες ερωτήσεις, ναι, ναι. Θέλετε να απαντήσετε απευθείας σε αυτό. Μα έγιναν δύο ερωτήσεις που δεν, στις οποίες δεν απαντήσαμε. Ναι, δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά συνέβη. Δεν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ε, απαντήσεις τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε μια ερώτηση που έκανε πριν από λίγο η κυρία Πρόεδρος και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς μπορεί η άμεση δημοκρατία στο ευρωπαϊκό επίπεδο να οδηγήσει στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το σκέφτηκα όπως ερχόμουν εδώ πέρα και νομίζω πως υπάρχει εδώ πέρα ένα δυναμικό το οποίο δεν έχουμε αναγνωρίσει γιατί δεν υπάρχει καμία εμπειρία. Η θεσμική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μοναδική στο πλαίσιο αυτό. και δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά βεβαίως πρέπει να πούμε πως για κάποιον αριθμό πολιτών υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουν βέτο κατά ενός ε, νόμου, ο οποίος δεν έχει τεθεί ενισχύ, αλλά έχει εγκριθεί και θεσπιστεί. Υπάρχει δηλαδή ε, για νόμους. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη ευκαιρία να φροντίσουμε εκ των προτέρων να μην προβάλλει κανείς βέτο, να μην ζητήσει κανείς δημοψήφισμα και εδώ πέρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή να υπάρξει μια διαδικασία διαμεσολάβησης έτσι ώστε να γίνουν να ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες αντιρρήσεις των πολιτών περισσότερο από ότι σήμερα για να μην υπάρχει όλη αυτή η δαμόκλειο σπάθη πάνω από την όλη διαδικασία ότι στο τέλος δηλαδή μπορεί να υποβληθεί ένα βέτο και υπάρχει απέναντι σε αυτό το βέτο μόνο η δυνατότητα να λάβει κανείς υπόψη ε, όλες αυτές τις αντιρρήσεις και αυτή είναι μεγάλη ε, ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω πως έτσι θα ενισχυθεί και θεσμικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα για το ερώτημα του κύριου Χέφνερ. Θεωρώ, για να είμαι σύντομος, για να είμαι σύντομη, πως τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας, τα οποία παρουσιάστηκαν, νομίζω πως μπορούμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Τι μας απαγορεύει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα με το να αναβάλουμε κάποια. Βεβαίως, εντάξει, είναι πολύ υποκειμενική η άποψή μου, αλλά θεωρώ πως ε, συγκεκριμένες καταστάσεις δείχνουν την ανάγκη των πολιτών να μιλήσουν και αυτοί. Ε, με το ίντερνετ, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε συζήτηση, υπάρχει άνοδο του κόμματο των ε, πειρατών, υπάρχει γενικώ ένα δημοκρατικό κύμα. Γιατί να μην αναγνωρίσουμε αυτή την ε, τάση για να ληφθούν υπόψη αυτές οι ανάγκες. Το άλλο ερώτημα, πώς η άμεση δημοκρατία μπορεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Πώς μπορεί να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Νομίζω πως είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να κατευθυνθεί, αλλά εμέσως η άμεση δημοκρατία θα μπορούσε να έχει κάποιες επιδράσεις. Στην ε, ελβετική εμπειρία, το ακούσαμε ήδη, έχουμε μια επίδραση αν θέλετε που ενώνει τους πολίτες, όχι μόνο την μιλάει κανεί με τους υπόλοιπους Ελβετούς συμπολίτε του, αλλά σημαντικό είναι επίσης το ότι τα όρια μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού δεν είναι έτσι μόνιμα. Και σε αυτό έχει ρόλο η άμεση δημοκρατία, παραδείγματο χάρη αναφέρατε το γλωσσικό σύνορο το ε, σύνορο το θρησκευτικό και βεβαίως ε, το σύνορο μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Αυτά βεβαίως ε, δεν είναι πάντα δεδομένα. Δεν σημαίνει πως κάποιος ο οποίος ζει στην πόλη έχει την ίδια θρησκεία και θα συμφωνεί πάντα με κάποιον στην ίδια κατάσταση. Είναι πάντα διαφορετικές οι σωματώσεις. Και δεν είναι βεβαίω πω κάποιοι είναι μονίμως σε μειονεκτική θέση. Κάθε πολίτης που έχει δικαίωμα ψήφου βρίσκεται μία φορά ε, σε μία ψηφοφορία ε, με τη μεριά των κερδισμένων, άλλη φορά με τη μεριά των χαμένων και νομίζω πως κάτι τέτοιο σε μια ευρωπαϊκή διάσταση θα ήταν ακόμη σημαντικότερο και θα είχε έτσι ένα αποτέλεσμα ενοποιητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, και εγώ να υπογραμμίσω ε, ορισμένα από αυτά που ελέγχθησαν. Δηλαδή, οποτεδήποτε υπάρχουν δικαιώματα ε, δημοψηφίσματο ή το δικαίωμα τη αρνησικυρία, τότε το σύστημα αντιδρά με την έννοια ότι προσπαθεί να παρεμποδίσει την άσκηση αυτού του δικαιώματο αρνησικυρία. Ένα από του καλύτερου ε, συνταγματολόγους ε, της Ελβετίας ε, είπε ότι και η ύπαρξη μόνο ενός δημοψηφίσματος οδηγεί στο να μπορούμε να επιτύχουμε αυτά που είναι τα πιο σημαντικά. Όχι όλα, αλλά τα πιο σημαντικά. σήμερα ήδη αναφέρθηκε ότι αν το σκεφτούμε λιγάκι προς τα κάτω, όπως είναι η πρωτοβουλία των πολιτών που επένεσε τόσο πολύ ο Μπρούνο, αυτό ε, δεν είναι γνήσιο δημοκρατικό στοιχείο όπως το εννοούμε εμείς. Γιατί ένα τέτοιο πρέπει να οδηγήσει σε δημοψήφισμα. Είναι υποβολή αίτηση προς εκείνους οι οποίοι έχουν σήμερα το μονοπόλιο του δικαιώματος ανάληψης πρωτοβουλίας, προς την Κομισιόν δηλαδή. Αν το συρρυκνώσουμε λιγάκι, το δικαίωμα κυρίες, αφορά ε, λίγους ανθρώπους στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό κοινό Κοινοβούλιο αλλά και σε όλους τους άλλους που, είναι, ε, που, που περιλαμβάνονται στην ε, νομοθετική εξουσία τους δίνει λοιπόν δυνατότητα στους ανθρώπους να ζητήσουν τη δεύτερη ανάγνωση. Οι εμπλεκόμενοι, οι υπουργοί, οι βουλευτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνοι που θίγονται άμεσα αλλά δεν ε, εκφράζονται. Και αυτό είναι η συμμετρική, συμμετρική αναλογία του δικαιώματος πρωτοβουλίας για δεύτερη ανάγνωση, χωρίς όμως να προκύψει δημοψήφισμα. Είναι, αν θέλετε, μία πολύ περιορισμένη επέκταση των συμμετοχικών δικαιωμάτων με στόχο οι ε, θεσμοί να ακούν όχι μόνο την άποψη των ομάδων πίσεων, αλλά και των υπολείπων ανθρώπων που δεν εκπροσωπούνται από αυτές τις ομάδες πίεσης. Γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα να ζητήσουν κάτι, κάτι που αλλιώς δεν θα το έκαναν αν είχαν την αίσθηση ότι θα τους αγνοούσαν. Και κάτι άλλο που νομίζω ότι μπορεί να ε, συμβάλλει στη συζήτηση. Πόνς ε, ήταν ένας Γερμανός καθηγητής που ε, μετανάστευσε στις ΗΠΑ και τον έλεγαν, τον αποκαλούσαν Mr. Deutsch. Αυτός λοιπόν ορίζει την εξουσία με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Είπε η εξουσία είναι το προνόμιο του να μην είσαι αναγκασμένος να μάθεις. Και αν είχε ακούσει εμάς, θα έλεγε, η εξουσία είναι το δικαίωμα του να μην είσαι να ακούσεις. Γιατί πριν μάθεις πρέπει να ακούσεις. Σε μία λοιπόν δημοκρατία, κανείς Μα πραγματικά κανένας πολίτης, κανένας θεσμός δεν πρέπει να έχει αυτή την εξουσία του να απορρίπτει τη μάθηση. Με αυτή την έννοια το να αναγκάζει κανείς να ακούσουν αυτοί που δεν θέλουν, ήδη αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό ακριβώς ε, συζητήσαμε όταν ε, μιλήσαμε για την ε, άμεση δημοκρατία. Όταν καλείται κανείς να σχεδιάσει το πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας. Δεν είναι όλοι ίσοι, αλλά η διαφορά δεν είναι όπως το γαλλικό σύστημα όπου ο ε, βασιλιάς επανήλθε από την πίσω πόρτα γιατί οι άνθρωποι είχαν ενοχές επειδή τον είχαν δολοφονήσει. Και τώρα, στην ερώτηση του Γκέραλτ, νομίζω ότι εκείνοι οι οποίοι συρρυκνώνουν τη δημοκρατία και την πολίτη, ε, δηλαδή λένε ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά τότε εντάξει συζητάμε, αυτοί δεν έχουν ποτέ καταλάβει την αξία της συζήτησης ή πιστεύουν ότι ο πολίτης είναι υπήκος. Και μόνο όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά έχει κανείς το χρόνο να τον ακούσει. Όμως να βρεθεί μια λύση ή μια ιδέα σε αντιπαράθεση με την άλλη πλευρά, αυτό φαίνεται δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, Για αλλιώ δεν θα το ξεχνούσαν. Και έτσι λοιπόν η κυρία Λίμπε είπε στην αρχή πολύ σωστά ότι κανένα, καμία χρονική στιγμή δεν ενδείκνεται τόσο πολύ όσο η κρίση για να αλλάξει ποιότητα. Γιατί η κρίση είναι η έκφραση αυτού ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο Γκράμψι είπε ότι όλοι ξέρουν ότι έτσι μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς να γίνει η αλλαγή. Αν λοιπόν δεν το ξέρουμε, καλύτερα να ακούμε, γιατί ίσως από κοινού να βρούμε κάτι. Ο Τέο λοιπόν αναφέρθηκε ε, στις κρίσεις ε, που στην ιστορία πάντα οδήγησαν σε δημοκρατία και είπε η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη αλλά δεν υπάρχει προτιμία να γίνει το επόμενο βήμα όπως έγινε στις ΗΠΑ Πολιτείες και στην Ελβετία, γιατί οι άνθρωποι ε, πήραν ξαφνικά την εξουσία στα χέρια τους και όχι οι φιλελεύθεροι. Αυτά όλα δεν γίνονται προαιρετικά, αλλά αν οι άνθρωποι κάτι κάνουν για να εισακουστούν, τότε εισακούονται. Εάν εμείς δεν ε, φοβούμαστε ότι δεν θα επανεκλεγούμε, τότε ακούμε τις επιθυμίες των ανθρώπων. Και ο φόβος αυτός ε, υπάρχει περισσότερο σε εκείνους που οφείλουν την εκλογή τους ανθρώπους. Και επίσης ε, ούτε η συντακτική συνέλευση αρκεί, γιατί αυτό αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά μπορούμε να οργανώσουμε, ε, αν θέλετε, μια συντακτική συνέλευση, χωρίς όμως νόημα. Αυτό σημαίνει ότι τον ξεφτιλίζουμε με την έννοια ότι η συντακτική συνέλευση διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Εγώ, ας πούμε, στην ε, Ελβετία, στην ε, Ζυρίχη, δύο φορές ε, βίωσα την τροποποίηση συντάγματος. Είμαστε σε ένα καντόνι που έχει συνηθίσει να αλλάζει το σύνταγμα. Εδώ όμως χρειάζεται περισσότερος χρόνος γιατί δεν το έχουν συνηθίσει και μάλιστα ακόμα δεν έχουν συζητήσει για τις ε, διάφορες ε, έννοιες που αποδίδουν οι διάφοροι λαοί στον όρο σύνταγμα. Αν όμως δεν το έχεις κάνει αυτό, δεν μπορείς να συμφωνήσεις ε, στο σύνταγμα η Αυστρία και αυτή αλλάζει συνεχώς το συνταγμά της χωρίς να το πάρουν χαμπάρι άνθρωποι ε, στην ε, Σουηδία κάθε 30 χρόνια όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία είναι κάπου στη μέση. Αυτή λοιπόν η συντακτική συνέλευση και αυτή η λέξη προέρχεται από την Αμερικανική ιστορία αυτή σημαίνει ε, μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση ανθρώπων που τους έχει ανατεθεί ακριβώς αυτό το έργο. Σήμερα το πρωί το θίξαμε. Ε, σε μια δημοκρατική ε, συνταγματική διαδικασία όπου όλοι στο τέλος ε, μπορούν να πούνε ναι ή όχι. Πρέπει κανείς να δείξει σε όλους ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του αυτά τα οποία λέγονται. Το 1995 με είχατε προσκαλέσει ήδη εδώ όταν έγινε κατανοητό ότι θα έπρεπε να ενταχθούν, να αφομοιωθούν και οι άνθρωποι και όχι μόνο οι λαοί. Αυτό όμως ήταν τότε καθαρά για το Θεατήν, ήταν βιτρίνα. Ε, τίποτα δεν έγινε, μεγάλη απογοήτευση και αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Όσον αφορά τώρα την ταυτότητα, ο Φρίσ είπε ότι την ταυτότητα δεν την κληρονομεί κανεί, κανείς, η ταυτότητα προκύπτει από την κοινή πράξη ε, και έμεσα όπως είπε προηγουμένως η κυρία Μπράουν. Ε, παθητικά όμως ε, χάνει κανείς την ταυτότητα. Ε, παθητικά δεν υπάρχει κοινή ταυτότητα. Γι' αυτό η αποκοινού πράξη είναι καθοριστική σημασίας. Και το τελευταίο θέμα. Υπάρχει λέξη δημοψήφισμα, το οποίο προφανώς έχει μια αρνητική χρειά, ακριβώς γιατί δεν έχουν αναλυθεί σωστά οι διάφορες εμπειρίες. Ο Τέο το είπε αυτό. Οι Γάλλοι χρειάστηκαν μισό χρόνο για να ε, καταλήξουν, να συμφωνήσουν ε, στη συντακτική συνέλευση. Και σε αυτή τη συζήτηση συνειδητοποίησαν πράγματα με τα οποία διαφωνούσαν. Τώρα λοιπόν καλείται κανείς ε, να αντιδράσει, υποβάλλει ένα νέο σχέδιο όπου δεν περιλαμβάνονται όλα αυτά που ήθελαν οι Γάλλοι και όχι μόνο οι Γάλλοι αλλά κανονικά όλοι οι Ευρωπαίοι. Αν δει κανεί λιγάκι την ιστορία τη Ευρωπαϊκή Συνταγματική Ιδέα, θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι πολύ πιο μεγάλη. Ε, τη δεκαετία του 50 στον πόλεμο ε, στις φυλακές των φασιστών όπου είχαν εγκλειστεί Ευρωπαίοι δημοκράτες και όπου συνέτασαν άρθρα με τα οποία έδειχναν πώς, ποια μορφή πρέπει να λάβει η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, ο Σπινέλη παραδείγματο χάρη, αυτά όλα τα κείμενα διέπονται από ε, ομοσπονδιακό πνεύμα με τον πολίτη και όχι κατά του πολίτη. Αυτά βέβαια τα εμπόδισε ο ψυχρός πόλεμος και η δυτική η Ευρώπη πλήρωσε λόγω του ψυχρού πολέμου ένα υψηλό τίμημα. Από την συνθήκη έγινε σύνταγμα και τελικά καταλήξαμε από την πολιτική να προκύψει η οικονομία. Στο τέλος λοιπόν του ψυχρού πολέμου υπήρξαν πολύ λίγοι όπως ε, και η Γερμανία οι οποίοι σκέφτηκαν ότι τώρα όμως πρέπει να καλύψουμε το κενό, αυτό που πριν από 30 χρόνια δεν ήταν δυνατόν, τελικά όμως δεν έγινε τίποτα. Προχώρησε βέβαια λογική, ε, προέκυψε το ευρώ χωρίς όμως θεμέλια, σαθρά θεμέλια και γι' αυτό πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Ούτε και η συνθήκη προχωράει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε θάρρος. Η συνθήκη σημαίνει ή ε, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του πολίτη. Η Γερμανία δεν είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Γαλλία, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτέ όλε αγωνίζονται με τον πολίτη, περιλαμβάνουν τον πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε το Σύνταγμα μαζί με τον πολίτη για την εμπέδωση τη έμεση και τη άμεση δημοκρατία. Σα ευχαριστούμε ο καθηγητή ε, Θα είμαι σύντομος ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ακούστηκε μεταξύ της κυρίας Λίμπερτ και του κύριου Χέφνερ. Ποια είναι η ποιότητα της διαβούλευσης και γιατί έχει σημασία αυτή. Πριν από 15 χρόνια εγώ είχα αναπτύξει μια θεωρία που ε, λέγαμε, που την ονομάζαμε διαβουλευτικός ε, υπερεθνικισμός αντί για ε, νομικός. Να δώσω ένα παράδειγμα φανταστείτε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα φάρμακο και θέλετε να μάθετε αν είναι ασφαλές. Είτε θα δείτε παραδείγματο χάρη το... τη γερμανική υπηρεσία αν το εγκρίνει και κάποια άλλα, π.χ. η δανέζικη υπηρεσία. Εμείς θεωρούσαμε πως ο πλουραλισμός αυτός είναι από μόνος του μία αξία γιατί έτσι υπάρχει η διαβούλευση. Οπότε το σκεφτικό εγώ και ο Γιώργεν κάναμε εμπειρική έρευνα, μιλήσαμε με ανθρώπους. Τόσο μην λιβανίζω και τα γένια μου. Αλλά το σκεπτικό του να λέμε θα περιμένουμε θα περιμένουμε να έχουμε ένα ενιαίο κράτος και μία ενιαία διοίκηση. Όχι, έχουμε κάτι άλλο και το κάτι άλλο αυτό είναι ε, κάτι το πλουραλιστικό. Εγώ σήμερα θα έλεγα πως πρέπει να συμπληρωθεί με στοιχεία ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης ε, ομάδων πολιτών και ενδιαφερομένων που μπαίνουν στη διαδικασία. Γιατί και πάλι δεν μπορούμε να περιμένουμε το ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος με τη μία διοίκηση κτλ. Χρειαζόμαστε αυτό το οποίο είπα, μία συνταγματοποίηση της συνεργασίας ε, των διαφόρων φορέων στην ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Τώρα από συνταγματοποίηση κακούγεται κάπως. Αν δείτε όμως τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δούμε αυτούς τους ειδικού να διαφωνούν και μετά στο τέλος λένε ε, εντάξει συμφωνούμε σε κάτι ας πούμε τουλάχιστον υπάρχει μια ποιότητα σε αυτή τη διαδικασία που είναι διαβούλευση ε, διαβούλευση βεβαίως δεν αποτελεί εγγύηση και η τάση δυστυχώς είναι ενάντια σε αυτό είναι να πάει σε μια αποκεντρωμένη υπηρεσία κτλ. Αλλά η αρχική ιδέα είναι πράγματι θέση, αντίθεση, επιχειρήματα και από αυτό να προκύψει μια συμφωνία. Μπορούν να συμφωνήσουν, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτά είχαμε πει τότε, βέβαια έχουν περάσει χρόνια από τότε. Πράγματι ήταν θετικό αυτό το οποίο είπατε γιατί δίνονται έτσι κίνητρα σε όλους και όλοι έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν νέες ιδέες και έτσι δημιουργούνται νέες ιδέες. Θα ήθελα να αντιδράσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φέφνερ. Είπε πως οι κρίσεις δημιουργούν και γεννάνε την αλλαγή. Για μένα οι κρίση ήταν πάντα ευκαιρία. Και το ερώτημα είναι πόσο σοβαρά παίρνουμε αυτή την ευκαιρία που μας προσφέρει η κρίση αυτή. Και βεβαίως πάντα ζητάμε βοήθεια όταν έχουμε προβλήματα, αλλά πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία εάν συνεχώς επιτηρούμε τη δημοκρατία και μόλις αισθανθούμε πως υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα πρέπει να δράσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη, υπάρχει μια σοβαρή κρίση και λέμε ναι εντάξει έχουμε περιορισμένα κονδύλια και με αυτά τα κονδύλια πρέπει να ξανασχεδιάσουμε την Ευρώπη. Οπότε προφανώς καταλήγουμε σε πολλά ερωτήματα και ανέφερε ο τέλος του 1995 που ήταν τελευταία φορά που ήρθε εδώ πέρα. Ελπίζω λοιπόν να είχε μια καλή ευκαιρία μια που ήρθε να μην μιλήσει μόνο στη δική μας επιτροπή αλλά και σε άλλες. Θεωρούμε πως ε, αυτές οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτή τη στιγμή θα έλεγα πως ζούμε στην καλύτερη δυνατή δημοκρατία. Έχουμε δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο, το, ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, αλλά το ερώτημα είναι ενδιαφέρεται ο κόσμος να το χρησιμοποιήσει αυτό ή όχι. Και ένα άλλο ερώτημα πρέπει να θέσουμε υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές συζητήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπάρχουν υπουργοί, πρωθυπουργοί που έρχονται στις Βρυξέλλες ε, και βεβαίως όταν έρχονται εδώ πέρα ε, είναι Ευρωπαίοι πολιτικοί και δρούν αναλόγως, μετά επιστρέφουν στη χώρα τους και με υπό άλλη ιδιότητα δρούν τελείως ε, διαφορετικά. Ως Ουγγαρέζα μπορώ να σας πω την εμπειρία μου για το πώς εγώ ζω την λεγόμενη Ουγγαρία στην ε, Ολλανδία. Το ερώτημα λοιπόν για το ποιος κυβερνάει την Ευρώπη ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ποιος κυβερνάει την Ευρώπη ξέρουν πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα πολύ ισχυρότερο από όσο ήταν στο παρελθόν χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και πώς θα επηρεάσουν τις καθημερινές τους ε, ζωές. Είναι πολλές αυτές οι ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους ε, συναδέλφους και τους ειδικούς. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, θέλω να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω τους παρόντους βουλευτές εάν έχουν ε, σχόλια ή ερωτήσεις ή ε, μπορούμε να ακούσουμε και ερωτήσεις από το κοινό ναι. Ο συναδελφός μου ο Λίβερ. Αλλά πρώτα απ' όλα σε ακούσουμε τους ειδικούς. Let me voice ε, a little doubt. Αν με επιτρέπετε να εκφράσω μια α, μικρή αμφιβολία με κάθε σεβασμό προς την πρόταση την οποία μας προτείνατε οι δυο σα. Νομίζω ότι η ενίσχυση των ε, δικαιωμάτων της λαϊκής αρνησικυρίας μπορούσε να είναι ενδεχομένως ε, σε αντίθεση με την ανάγκη να προταθούν αλλαγή, αλλαγές και στην επίλυση των εμφανιζόμενων προβλημάτων. Αν δηλαδή το ΒΕΤΟ βοηθήσει να ενισχυθεί το status quo, τι να σας πω. Φυσικά Πολλά μπορεί κανείς να πει υπέρ, αλλά εγώ θα ήμουν υπέρ της εκμετάλλευσης του δημιουργικού δυναμικού των πρωτοβουλειών που έχουν ως ε, στόχο την επίλυση προβλημάτων, νέο τρόπο διατύπωσης προτάσεων. Να βοηθήσουμε λοιπόν να αναπτυχθεί αυτό το δημιουργικό δυναμικό για την επίλυση των προβλημάτων ε, μέσω της δημοκρατίας της διαδικασίας. Input democracy. Έχετε εσείς κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, ε, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να βρούμε το θάρρος ε, κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Και αν ξεκινήσουμε, βεβαίω και υπάρχει ο κίνδυνος ε, οι άνθρωποι να επιθυμούν κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε εμείς. Όμως η πρόοδος τους ε, θα πρέπει δυστυχώς ε, να ξέρουμε ότι θα είναι ε, σποραδική, πολύ περιορισμένη, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει νομιμοποίηση και συνένεση. Έτσι και αλλιώς στη θεωρία ποτέ δεν είναι κατάλληλη στιγμή, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από τη στιγμή ε, της κρίσης. Τα τελευταία 30 χρόνια η αλωτρίωση ε, οξύνθηκε τόσο πολύ που οι άνθρωποι πλέον αισθάνονται δυσάρεστα και πρέπει να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε αυτούς τους ε, αλωτριωμένους να τους επανεντάξουμε. Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα πώς μπορεί κανείς ε, να προσπαθήσει γι' αυτό το αποτέλεσμα και όχι το αν θα προσπαθήσει. Και βεβαίως ε, δεν υποτιμώ τις προσπάθειες που είναι απαραίτητες, αλλά ειδικά τώρα είναι σαφές ότι το κράτος έθνος δεν είναι πλέον σε θέση να επισκευάσει κάτι. Χρειάζεται την Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί η Ευρώπη να γυρίσει την πλάτη στους πολίτες. επειδή μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση. Αν δύο από εσάς θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, ερώτηση, δεν ξέρω. Πραγματικά. Ε, έχετε τη δυνατότητα κι εσείς να σχολιάσετε. Restart or renew, ε, you have to be brave enough. Φυσικά ε, το θέμα είναι, είμαστε αρκετά γενναίοι ε, για να κερδίσουμε. Βέβαια, άμα δεν αγωνιστούμε δεν πρόκειται και να κερδίσουμε ούτως ή άλλως. Και είναι μια τέτοια περίοδος αυτή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για την Ουγγαρία, η ισότητα των δύο φίλων. Ε, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Είχαμε στο παρελθόν κάποια προβλήματα, τώρα ξαναβλέπουμε να υποχωρούν ίσως κάποια δικαιώματα, υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν προβλήματα με, ιδίως με επίκεντρο τη βία και έγιναν κάποιες συζητήσεις ε, και στο κοινοβούλιο και είπε κάποιος, αν κάποιος έχει δύο, τρία, τέσσερα, πέντε παιδιά, είναι εγγυημένο ότι δεν υπάρχει βία στην οικογένεια και η συζήτηση βέβαια έγινε στην Ολομέλεια γιατί δεν ήταν γενναία για να βάλουν ε, το θέμα αυτό πιο νωρί στην ημερήσια διάταξη. Και άρχισαν αντιδράσεις ε, στην Ουγγαρία, τώρα κινούνται κάπως τα πράγματα. Και έχει ξεκινήσει και μάλιστα κράτησε ένα χρόνο και η συζήτηση για την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών ε, στα διοικητικά συμβουλία. Ε, οι υπουργοί από το Συμβούλιο λένε τώρα ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα των ποσοστώσεων και ούτε καν καταδέχουν να διαβάσουν το έγγραφο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχει διανεμηθεί στην, ε, εσωτερικά στην Κομισιόν το, το, το θέμα, έχει αρχίσει συζήτηση. Είναι απαράδεκτο λοιπόν κατά την άποψή μου το Συμβούλιο Αντί να καταλαβαίνει τι γίνεται, να βλέπει τι έγινε και κατά το παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να κάνει αυτά που κάνει. Τρία ψηφίσματα ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Και είχαμε και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο υπέρ τη άποψη ότι χρειαζόμαστε περισσότερε γυναίκε. Και πολλοί υποστήριξαν βέβαια ότι άμα έχουμε μεγαλύτερη γυναική εκπροσώπηση μπορεί να μειωθεί και η Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, αλλά τέλος πάντων σίγουρα αξίζει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες ούτως ή άλλως. Θα στείλουμε μια ανοιχτή επιστολή στου υπουργούς και θα τους ρωτήσουμε πώς μπορεί να είστε τόσο γενναίοι και να λαμβάνετε αποφάσεις χωρίς καν να έχετε μελετήσει ούτε καν διαβάσει το έγγραφο. Βλέπω την κυρία Ρενάρντα από την Κομισιόν, δεν είδα κάποιον άλλο να θέλει το λόγο. Κυρία μου, σας καλωσορίζω και θέλω να κάνετε και κάποια σχόλια, όχι μόνο στο δικό μου το τελευταίο σχόλιο, ε, αλλά και να σχολιάσετε ή να πείτε οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Έχετε τώρα την ευκαιρία να το κάνετε. Εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια ακρόαση. Σήμερα το πρωί οι συνάδελφοί μου που εργάζονται πάνω στο θέμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ε, πρόσεξαν. Ε, άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον όλα αυτά που ακούστηκαν και από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Γιούστε, οι συναδελφοί μου. Όλοι μαζί πιστεύω ότι θα μελετήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα συζητήσατε σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της Κομισιόν. So then we should recommend a type of trialogue on this issue because I believe... Άρα να, να προτείνουμε να γίνει τριμερής διάλογος για αυτά τα θέματα. Καλό θα ήταν. Είναι εδώ και επικεφάλη τη ε, γραμματεία και φαντάζομαι θα διαβιβάσει στον πρόεδρο Καζίνη την πρόταση αυτή. Υπήρξε ένα ερώτημα από εσά να μα ε, πείτε και ποιο είστε, από ποια χώρα κατάγεστε. Και η κυρία μετά θα μιλήσει. Ντόναλντ Μπράναγκαν, λέγομαι, είμαι από την Ιρλανδία. Δεν εκπροσωπώ κάποιον άλλον πέραν του εαυτού μου εδώ σήμερα. Νομίζω ότι κάποιος ε, ευρωβουλευτής έκανε ε, ορισμένα σχόλια για την Ιρλανδία που θα έπρεπε να τα διορθώσω. Μόνο ένα ε, ψήφισμα είχαμε για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο στη χώρα μου και πέρασε. Είχαμε δύο όμως δημοψήφισματα για τη συνθήκη της Νίκιας και τη συνθήκη της Λισαβόνας που την πρώτη φορά και οι δύο είχαν απορριφθεί. Είχαμε δηλαδή δύο διπλά, όχι τρία διπλά δημοψηφίσματα. Κάποιοι λένε ότι είναι κατά της εξαγωγής δημοψηφισμάτων για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και πολύ σωστά. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί πλέον που μπαίνουν ε, στη δεξαγωγή των ε, δημοψηφισμάτων. Εμείς δεν έχουμε στην Ιρλανδία συνταγματικό δικαστήριο, έχουμε ένα όμως ανώτατο δικαστήριο, το οποίο επέβαλε κάποιους περιορισμούς, είναι το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει για συνταγματικά ζητήματα και ετέφει το εξή θέμα, σε ποιο βαθμό μπορεί η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε, ε, οποιοδήποτε δημοψήφισμα ε, και αυτό ε, το απέρριψε το δικαστήριο. Δεν μπορεί δεν μπορεί να, να το κάνει αυτό. Και τώρα ποια είναι η στάθμισή του ναι του όχι και πόσος χρόνος θα δίνεται για τις δύο πλευρές Όλα αυτά συζητήθηκαν, πάντως κάποιοι τάχθηκαν υπέρ, ε, μάλλον κατά, γιατί παλαιότερα είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να μιλήσουν. Μια ερώτηση προς το πάνελ, δεν ξέρω αν είναι αργά, προς τη δόκτωρα Λίμπερτη, πρώτη μου ερώτηση. Η άμεση δημοκρατία σε ποιο βαθμό προάγει και προωθεί την διαβουλευτική δημοκρατία, που ελπίζω να το κάνει. Προς τον δόκτωρα Γκρός, το ερώτημά μου είναι αν στα πέντε σημεία ε, της δικής σας ε, άποψης για την άμεση δημοκρατία. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εντός ε, του οποίου θα πρέπει τα αποτελέσματα ακριβώς αυτής της εφαρμογής της άμεσης δημοκρατίας είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο να υλοποιούνται και προς την ε, κυρία Μπράουν ε, Βίντερ οι ηλεκτρονικές υπογραφές σε ποιο βαθμό τώρα ε, που μπαίνουν στο ομοσπονδιακό επίπεδο στην Ελβετία, έχω ε, διαβάσει κάποια πράγματα, ε, υπάρχουν κάποιες εμπειρίες σε επίπεδο καντονιού και χαμηλότερο. Τι θα γίνει όμως με το εθνικό επίπεδο. Η πρόοδος έχουμε και μια ερώτηση από τα αριστερά και άλλες δύο από τα δεξιά. Και οι συνάδελφοί μου θα απαντήσουν και μετά θα κάνουμε και μια σύνοψη. Είμαι Είμαι φυσικό και με την πληροφορική και είμαι εδώ πολλά χρόνια. Έχω δει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Αυτή η πρόταση με ενθουσιάζει. Είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο ε, όμως αυτή η πρωτοβουλία. Όχι, είναι ένα ε, μια προσέγγιση κατά την άποψή μου. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό δημοψήφισμα και το πρώτο θα πρέπει να αφορά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα κατά την άποψή μου. Για να ξαναξεκινήσει αυτή η διαδικασία μέσω του δημοψηφίσματος του Ευρωπαϊκού. Εγώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που θα πρέπει να έχει τις εξουσίες για να ζητήσει ή να δρομολογήσει ένα ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Και νομίζω ότι αυτό το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα μπορεί να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες όπου η λεγόμενη δημοκρατία υπάρχει. Ε, Παραδείγματος χάρη πρώην ε, κομμουνιστικές χώρες που έρχονται εδώ οι επικεφαλείς αυτών των χωρών, λένε το ένα και μετά όπως είπατε πάνε στις χώρες τους και κάνουν κάτι εντελώ διαφορετικό και φοβούνται τα δημοψηφίσματα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και προβλήματα. Για μένα λοιπόν και αυτό που προτείνω είναι να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μπορεί να καθιερωθεί τάχιστα το ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Τελευταία μου πρόταση είναι ότι ένα ευρωπαϊκό δημοψήφισμα, τώρα δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε να το οργανώσετε, αλλά και κατ' εμέ πρέπει ένα ευρωπαϊκό δημοψήφισμα να αναφέρεται σε ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκού συντάγματος, αλλά αν αναφέρεται και με πάρα πολύ επίκαιρα φλέγοντα προβλήματα, όπως είναι η οικονομική κρίση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία. Τι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι σχετικά. Πρώτος, άρα τελευταίο ερώτημα, εσείς εκεί αριστερά. Μια μικρή παρατήρηση. σε μήλου, φλέγομαι και δουλεύω για μια βελγική ΜΚΟ για την ε, ένταξη. Ε, συμμετοχή, συμμετοχική δημοκρατία. Δεν ξέρω, γνωρίζετε ότι έχουμε 20 εκατομμύρια μετανάστευση και θέλουμε ε, να ακουστεί και η δική μας φωνή στην Ευρώπη. θεωρητικά λέμε ότι πρέπει και λειτουργεί πολύ καλά, αλλά εγώ προσωπικά βλέπω να υπάρχουν δυσκολίες. Αν εγώ γράψω ένα email, μια επιστολή στο όνομά μου και αντίστοιχα ε, έχω ακούσει από μουσουλμάνους ε, ε, συναδέλφους ότι είναι δύσκολο να μας απαντήσουν. Δύο-τρεις ε, αν έχουν απαντήσει. Και έτσι πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς. Φυσικά και πρέπει να είμαστε ισότιμα μέλη της κοινωνίας. όσοι είναι εδώ στην αίθουσα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι υπέρ. Αλλά ξέρετε, στην κοινωνία υπάρχουν. Ε, ε πραγματικά υπάρχει χάσμα αυτή τη στιγμή μεταξύ των ε, αλλουδαπών και των ε, κατοίκων της χώρας. Και είστε, και ε, είσαστε και το... Ήσασταν ανησυχητέ για πολύ δύσκολο θέμα της Τσετσενίας. Σας ευχαριστώ. Ε, η διασπορά των Τσετσένων εδώ, τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, θα βιώσουν τη δημοκρατική εμπειρία και θα μεταλαμπαδεύσουν, ελπίζουμε, και στην ε, δημοκρατική κοινωνία εκεί αυτά, τις εμπειρίες τους αυτές. Ο πρόεδρος πράγματι. Ε, το θέμα είναι αν μπορεί να ακουστεί η φωνή σας είπατε δύο στις δέκα φορές, σας ακούν τέλος πάντων, δεν είναι... Δεν αρκεί αυτό. Ακούσαμε και κάποια σχόλια. Μπορεί να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που ετέθησαν. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πράγματι πρέπει πρώτα να σας ακούσουμε και μετά να αποφασίσουμε μαζί σας τι θα κάνουμε μετά. Και νομίζω ότι το ίδιο είπαν λίγο πολύ και όλοι η συνάδελφοι από το πάνελ ότι ναι, χρειάζεται μεγαλύτερη ε, αντιπροσώπευση, συμμετοχή, περισσότερη δημοκρατία. Αλλά πώς θα το πετύχουμε. Και νομίζω ότι εμείς ε, όλοι πιστεύουμε στο διάλογο, είμαστε όλοι αγωνιστές, ε, θέλουμε δικαιώματα για τους μετανάστες, για τα άτομα με αναπήρεια και το καθεξής. Όλοι είμαστε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον είμαι πεπισμένη φιλοευρωπαίστρια και σίγουρα θέλουμε να κάνουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, να παρακαλέσω τώρα τους ε, συναδέλφους του πάνελ να κάνουν ε, τις καταληκτικές τους παρατηρήσεις και θέλω να ευχαριστήσω και το κρατήριο τις ερωτήσεις του. The Irish experience... Η εμπειρία από τα Ιρλανδικά δημοψηφίσματα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσον αφορά το εάν και πώς μπορούμε να έχουμε το όραμα κάποια μέρα ενός πανευρωπαϊκού δημοψηφίσματος. Τρία ζητήματα λοιπόν υπάρχουν. Το ένα είναι η διαστρέβλωση της ε, συζήτησης λόγω των οικονομικών συμφερόντων. Υπήρχε και μία εκστρατεία υπέρ του όχι που είχε ε, χρηματοδοτηθεί αδρά στο πρώτο δημοψήφισμα. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, ε, που δεν αφορά μόνο την Ιρλανδία, αλλά οποιοδήποτε διποψήφισμα επικύρωσης που είχαμε στη Γαλλία, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, για την συνταγματική τότε συνθήκη, ο ρόλος των ΜΜΕ. Και από το Λάκεν στη Λισαβόνα κάναμε μία συγκριτική ανάλυση για τα ΜΜΕ, είδαμε το πλαίσιο, τα επιχειρήματα το πώς ε, έβλεπαν τη συζήτηση στα παλιά και νέα κρατημέλη. Είδαμε πολλές ε, διαφορές, πολλές ελλείψεις σε κάποια ΜΜΕ και βεβαίω δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον ρόλο των ε, ΜΜΕ και στην ελβετική εμπειρία. Ο Χανς Φέτερ Κρίζη νομίζω ένας πολιτικός επιστήμονας από τη Ζηρίχη που είναι τώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας κάνει τέτοια έρευνα πώς ε, να λάβουμε υπόψη τα ΜΜΕ που είναι δημόσια, ιδιωτικά, μεικτά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη το τρίτον που αφορά μια πρόταση που δεν έχει συζητηθεί, δηλαδή τι γίνεται με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών οι εθνικές, ε, υπερεθνικοί, υπερεθνικοί οργανισμοί, ΜΚΟ κτλ. Δεν μιλάω εδώ πέρα για ε, οικονομικά συμφέροντα, αλλά διάφορα συμφέροντα. Πρέπει να φροντίσουμε για να αντισταθμίσουμε τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα σε αυτές τις ε, εκστρατείες για τα δημοψηφίσματα και τη διαστρέβλωση που υπάρχει πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και να προετοιμάσουμε το έδαφος για την ενίσχυση των ΜΚΟ για να ζωθεί η πρόσβαση για να υπάρξουν διαβουλευτικά συνενετικά συνέδρια που μπορεί να γίνουν πριν από τρεις μήνες ε, από ένα τέτοιο δημοψήφισμα για να υπάρχει έντονη συζήτηση με τέτοια διαβουλευτικά συνενετικά συνέδρια που θα μεταδίδονται ευρέως. Concerning the Irish question, όσον αφορά το θέμα της ε, Ιρλανδίας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να δώσουμε μια γενική φύσεως απάντηση, γιατί εξαρτάται από το τι θέλει κανείς να αλλάξει. Μερικές φορές ε, αποφασίζει κανείς κάτι Κυριακή και τη Δευτέρα εφαρμόζεται και άλλες φορές είναι συνταγματικός νόμος, η συνταγματική διάταξη που χρειάζεται νόμο και όλα τα υπόλοιπα και μερικές φορές πρόκειται για μια συνεχή πρόκληση ε, που ποτέ κανείς δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Δεν μπορεί ε, να θέσει κανείς ένα χρονοδιάγραμμα που να ισχύει για όλα τα δημοψηφίσματα. Κοιτάξτε, κατά τα άλλα, θέλω να σας πω ότι αναφερθήκατε σε μια έκθεση που για να βρει κανείς ένα δημοκρατικό χαρακτήρα σε ένα δημοψήφισμα, όλοι θα απογοητευτούν μετά από το δημοψήφισμα. Πρέπει να υπάρξει όμως ε, μία διαδοχή, αν θέλετε. Άρα θα πρέπει να τεθούν και νομικά ζητήματα συνταγματικού δικαίου, αλλά και ουσιώδη θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με την πραγματικότητα. Αυτό θα κινητοποιήσει τον κόσμο. Θα πρέπει δηλαδή ο κόσμος να αναγνωρίσει ότι αντιμετωπίζονται προβλήματα της καθημερινότητάς του. Αυτό είναι η δημοκρατική κουλτούρα, η δημοκρατική νοοτροπία που χρειαζόμαστε. Και επίσης ε, πολύ ευγενικά ήταν αυτά που είπατε για την Τσετσενία. Με όλο πως τον Ταγκεστάν πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας σήμερα. Εκεί ε, στο Βιβία μπορεί ε, τα πράγματα εκεί να μην είναι και βέβαια και τόσο ξέθαρα. Τέλος πάντων πάρα πολύ ξεχασμένοι, πολύ λησμονημένοι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό επίση και στην Ελβετία πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν την άμεση δημοκρατία που υπάρχει. Και χρειάζονται πολιτικά δικαιώματα που να καλύπτουν ευρύτερο στρώμα της κοινωνίας. Ίσως να είναι καλύτερα ε, το γαλλικό τμήμα της Ελβετίας παρά το γερμανικό. Γιατί υπάρχουν με την ψηφοφορία, με τις εκλογές για την πρώτη Βουλή και τη δεύτερη υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια προβλήματα. Σίγουρα δεν είναι υποδειγματικά τα πράγματα και στην Ελβετία πάντα, αλλά μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τη δεκαετία του 1860 νομίζω ότι καταφέραμε να αξιοποιήσουμε πολλά από τα επιτεύγματα αυτής της Επανάστασης. Το θέμα ότι αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δεν είναι πλεονέκτημα του Ελβετού υπηκόου. Το θέμα είναι να υπάρξει επαρκή προστασία των βασικών δικαιωμάτων, ώστε δεν, να μην έχουμε ε, την τυραννία της πλειοψηφίας κατά της πλειοψηφίας και αυτό να θεωρείται άμεση δημοκρατία. ίσως σε άλλες χώρες να λαμβάνονται, να ε, είναι καλύτερες οι διαδικασίες από τη στην Ελβετία. Επιτρέπετε. Ε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας για την ηλεκτρονική υπογραφή και την ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών. Η Ελβετία έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία με τηλεψηφοφορία ε, και με τον υπολογιστή έξω από τα εκλογικά τμήματα μέσω διαδικτύου όμως η Ελβετία δεν έχει καμία εμπειρία με ηλεκτρονική υπογραφή για δημοψηφίσματα ή πρωτοβουλίες πολιτών κτλ. Γιατί η Ελβετία έχει πάνω από 2.000 δήμους και κάθε δήμος τηρεί δικό του εκλογικό κατάλογο και δεν υπάρχει ένας ενιαίος πανεθνικός. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο τονίζω πως είναι τόσο σημαντικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο να λυθεί το ζήτημα της υποδομής πριν ε, εισαχθούν τέτοια μέσα. Και πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τυποποιημένοι αν όχι εναρμονισμένοι εκλογικοί κατάλογοι για να ελέγχει, να, να υπάρχει δυνατότητα να, ελεγχθεί αν κάποιος ε, έχει δικαίωμα να υπογράψει και να ψηφίσει ή όχι. Και δεν έχουμε λοιπόν τέτοια εμπειρία εμείς. Σας ευχαριστώ κύριε Χέφνα. Ναι. Τέλος. Δεν θέλω να κάνω καμία ερώτηση, απλά να αναφέρω κάποιες σκέψεις. Äh, Πρώτα απ' όλα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες για την έξοχη αυτή ακρόαση. Θεωρώ πως Όλοι το ξέρουμε αυτό όπως κάνει τεράστια διαφορά στην αυτοεκτίμησή μου στο τι αποφάσεις παίρνω, στο πώς είμαι σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, το εάν ε, αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως ε, έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αποφασίσει μόνος του για κάποια πράγματα ή εάν μονίμως θεωρώ εαυτόν ε, υπόδουλο της, ε, των αποφάσεων των άλλων. Γιατί αν κάποιος ε, αισθάνεται ότι υποτάσσεται στη θέληση των άλλων, αυξάνεται η οργή και κάποια φορά οδηγεί στη βία και αντιστρόφως, εάν κάποιος ε, θεωρεί ότι τον παίρνουν σοβαρά και συμμετέχει και τον ρωτάνε, μπορεί να συμβιβαστεί με αποφάσεις που δεν θα λάμπανε ο ίδιος, αλλά τιμά το ότι και αυτός συμμετείχε στη διαμόρφωση και αποδέχεται άρα το αποτέλεσμα. Αυτό για μένα είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε αυτό το μυστικό στην, στην πολιτική, γιατί πρέπει να το πω ανοιχτά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο δυσάρεστη δουλειά από αυτή του πολιτικού. Στη Γερμανία τουλάχιστον υπάρχει κάθε έτος ε, μια δημοσκόπηση για την εκτίμηση που απολαμβάνουν ε, τα διάφορα επαγγέλματα. Η πολιτική είναι κάτω από τους πολιτές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Αντιλαμβάνεστε. Δουλεύουμε εδώ πέρα μέρα νύχτα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το κοινό καλό και ταυτόχρονα μας επιτίθενται από παντού γιατί οι πολίτες έχουν την αίσθηση πως ε, με ποιο δικαίωμα εσείς ε, κρίνετε το τι θέλουμε εμείς. Και ειλικρινά δεν το ξέρουμε. Όχι μόνο εδώ μέσα, σε αυτό το κοινοβούλιο, αλλά επειδή ήμουν βουλευτής και σε άλλα κοινοβούλια, πρέπει να πω πως εδώ είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι παραδείγμα τους χάρη στη Γερμανική ε, Ομοσπονδιακή Βουλή. Είμαστε πολύ μακριά από τον πολίτη οι πολίτες είναι πολύ μακριά από αυτά τα θεσμικά όργανα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και καμιά φορά αισθάνομαι ότι μιλάω από... όχι απλά από καθέδρας, αλλά πάρα πολύ απομακρυσμένος από τον λαό. Και δεν υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα να συζητήσουμε όλες τις εναλλακτικές και από την άλλη οι πολίτες λένε «Μα εμείς δεν, μιλάμε ποτέ, δεν, δεν ακούγει τη φωνή μας». Οπότε... Είπαν και οι συνάδελφοι ούτως ή άλλως πολύ πιο αναλυτικά από μένα. Η Ευρώπη είναι συνθήκες οποίες υπέγραψαν οι κυβερνήσεις εξ ονόματος των λαών. Οπότε το θεμέλιο αυτής της Ευρώπης χτίστηκε χωρίς τους λαούς. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε το κοινοβούλιο και αποκτά επιρροή, αλλά εξακολουθεί αυτή η Ευρώπη να είναι μια Ευρώπη η οποία κατά βάση είναι μια διακυβερνητική σύμβαση, μια συνθήκη μεταξύ κυβερνήσεων και όχι ανθρώπων. Και αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πως στο λίκνο αυτό, αν θέλετε, της Ευρώπης θα έπρεπε να βρίσκονται οι πολίτες και όχι τα κράτη. Και πραγματικά, εάν κάτι με, με με απογοητεύει είναι η θρηλυκή μας ανικανότητα να διδαχτούμε από τα λάθη μας. Εγώ το καλοκαίρι ήμουν στις ΗΠΑ ε, και μετά με προσκάλεσε ο Αμερικανός πρόξενος στο Μόναχο να του πω τις παρατηρήσεις μου στις ΗΠΑ και τι έμαθα στην πατρίδα της ε, δημοκρατίας ε, και πώς βλέπω την Αμερικανική δημοκρατία κτλ. και σκέφτηκα πως όταν κάποιος κάνει κάτι πρώτος δεν έχει ίσως την καλύτερη λύση, ίσως οι άλλοι που έρχονται μετά ε, σκέφτεται λογικότερα. Π.χ. δεν θα είχαμε τους εκλέκτορες που έχουν οι Αμερικανοί δεν μπορεί πριν από 200 χρόνια όταν ιδρύθηκε η χώρα να έχει νόημα να στέλνουν τους εκλέκτορες με το άλογο στην πρωτεύουσα και να λένε αυτή ήταν η απόφαση της πολιτείας. Ε τώρα είναι μπουρδες αυτά τα πράγματα. Αμέσως φαίνεται τι ψήφισαν στο Τέξας και στο Wisconsin και στα λοιπά. Δηλαδή το να μπαίνουν στη μέση οι εκλέκτορες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό πρόεδρο. Βεβαίω δεν θα καταργηθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα καταργηθεί το σύστημα. Δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. Και ε, αυτά με απογοητεύουν και βρίσκω πάρα πολλά τέτοια στην Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή κάποια θεμέλια που πλέον δεν αντέχουν από αυτά τα, πολλά από αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο. Μιλάμε για οικονομική διακυβέρνηση. Δεν καλύπτεται από το... Δεν, δεν βασίζεται και νομικά πουθενά στην Ευρώπη. Δηλαδή το οικοδόμημα αυτό έχει ξεφύγει τελώ και γίνεται όλο και πιο ασταθέ. Πρέπει να επεκταθούν τα θεμέλια κάποια στιγμή. Να πούμε χρειαζόμαστε ευρύτερα θεμέλια για να μπορούν να φέρουν αυτό το οποίο χτίζουμε. Για να έχουμε μια κοινή παραδείγματο χάρη ευθύνη στην Ευρώπη και για να υπάρχουν και υγιή δημοσιοοικονομικά αλλά και αλληλεγγύη παραδείγματο χάρη. Γιατί λένε οι Γερμανοί, μα γιατί η Μέρκελ δεν κάνει περισσότερα για τα συμφέροντά μα, Οι Γερμανοί λένε, οι Έλληνες λένε γιατί μας τα κάνουν όλα αυτά οι Γερμανοί. Δηλαδή, αν θα ήθελα κάτι εγώ, θα ήθελα μια Ευρωπαϊκή Συνέλευση. Η κρίση νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό. Εδώ πέρα συμφωνώ απολύτως. Που θα έχει ως αποστολή να φτιάξει νέα θεμέλια για την Ευρώπη, δημοκρατικά θεμέλια για μια Ευρώπη των πολιτών και θεμέλια για μια Ευρώπη που μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κρίση, γιατί δεν είναι κρίση ε, όσον αφορά τις ε, συναλλαγές των τραπεζών. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα. Δεν φτιάξαμε τους σωστούς κανόνες για να εμποδίσουμε ορισμένα πράγματα να συμβούν και τώρα ρίχνουμε συνέχεια λεφτά, αλλά η αιτία του προβλήματος δεν έχει παραμεριστεί και πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Εκεί πέρα λοιπόν είναι η αποστολή μας και αν συνεισφέραμε εμεί σήμερα, ε, έστω και ελάχιστα, εμείς δηλαδή, ή εκπρόσωποι των πολιτών. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για τους εαυτούς μας, είμαστε για να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες. Εάν Καταφέραμε λοιπόν να μην φοβόμαστε τους πολίτες και τη συμμετοχή τους, αλλά να τους δούμε ως συνεταίρους μας και τελικά ως κυρίαρχο λαό, να φτιάξουμε μια Ευρώπη με τους πολίτες, για τους πολίτες, νομίζω πως ήταν επιτυχής η σημερινή ακρόαση. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τη Ζήτα Γκουρμάη, τον Κάρλο Καζίνη που διευθύνει εξαιρετικά τη συζήτηση και ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ομιλητές μας που ε, απάντησαν εξαιρετικά σε όλες τις δύσκολες και χαζές ερωτήσεις που ακούστηκαν και την Κομισιόν και το Συμβούλιο που ήταν εδώ πέρα από την αρχή μέχρι το τέλος και παρακολουθούσαν και όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε ως πρόεδρος θέλω και εγώ να αναφέρω έξι σημεία θέλω να αναφέρω ε, το κρυφό δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει μία μοναδική ε, θεσμική θέση και πράγματι έχει μία μοναδική θέση, να, ένα μοναδικό ρόλο να παίξει και θα συνεχίσει η σημασία όταν να αυξάνεται τα επόμενα έτη, όχι μόνο λόγω των θεσμικών αλλαγών της συνθήκης Λισαβόνας, αλλά και λόγω της θέσης του ως ε, θεσμικό όργανο, το οποίο είναι ερετό άμεσα χρειάζεται περισσότερη ορατότητα. Αν θέλετε, πράγματι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα προνόμια του και βεβαίω μεγαλύτερη διαφάνεια. Το δεύτερον, Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια εντό των θεσμικών οργάνων και περισσότερη γνώση για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλοί πολίτε δεν γνωρίζουν ακόμα το τι γίνεται από τους εθνικούς πολιτικούς και ειδικά τους ευρωσκεπτικιστές. Ε, το επόμενο σημείο, το να ακούμε τους πολίτες, ε, πράγματι η εξουσία είναι το προνόμιο να μην χρειάζεται κανείς να ακούει και να μάθει. Πράγματι, τέταρτον για τα σχόλια ενός ε, ομιλητή για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και το ότι δεν είναι άμεση δημοκρατία και βεβαίω το ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα να ζητήσει κανεί δεύτερη ανάγνωση. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι εργαλείο συμμετοχική δημοκρατία, όχι άμεση δημοκρατία. Είναι δύσκολο αυτό η άμεση δημοκρατία σε τόσο μεγάλη ε, έκταση όπω ε, αυτή που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαφορετικά τα πράγματα λοιπόν από, το Ευρω... από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και επιπλέον, όπω είδαμε και με την Άκτα, αν οι πολίτε αρχίζουν να κινητοποιούνται, η φωνή του ακούγεται. Πέμπτον, η δημοκρατική συμμετοχή που προκύπτει από τα, το εκλογικό δικαίωμα δεν μπορεί να επιβάλλεται στους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καθημερινή ζωή του πολίτη και βεβαίως πρέπει να πουλήσουμε το προϊόν. Το προϊόν λέγεται Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν ξεκάθαρες πληροφορίες για το τι μπορούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Και βέβαιω η κρίση που μπορεί να οδηγήσει τη δημοκρατία σε νέο επίπεδο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο και πάλι βεβαίω θα αναφερθώ σε έναν ομιλητή μα. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προχωρούσε στις κρίσεις. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια κρίση άνευ προηγουμένου και επιπλέον οι απαντήσεις στην κρίση, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ε, έλαβαν χώρα σε κλειστές συναντήσεις Οπότε πρέπει και εμείς να ασκήσουμε κριτική στους εαυτούς μας. Λοιπόν, πριν κλείσουμε εδώ πέρα, Πριν λοιπόν σας ευχαριστήσω για την εμπειρία και τις ιδέες που μας μεταδώσατε, τώρα θα μιλήσω την ουγγρική, την μητρική μου γλώσσα. Η επόμενη λοιπόν συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 4 Οκτωβρίου 2012, 9 με 12.30 και μετά το απόγευμα 3 με 6 και 30 θα είναι ένα εργαστήριο την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Και μετά την 8η ε, Οκτωβρίου όλη μέρα και 9η Οκτωβρίου μόνο το πρωί, 9 με 12.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας διαβεβαιώ πως θα ενημερώσω τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, για να διαβιβάσει τις προτάσεις αυτές στην διάσκεψη των πρόεδρων. Τη δε περασμένη Παρασκευή Είχα την τιμή να παραβρεθώ σε μια συνάντηση με τον κύριο Γκρός ως πρόεδρος ε, των, της οργάνωσης γυναικών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ε, και έτσι μιλήσαμε για την οικοδόμηση ενός δικτύου γιατί είναι σημαντικό και για εμάς ε, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το τι είναι η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ